Αγαπητοί συνάδελφοι. Uh, um, Θα ήθελα να σας καλωσορίσω και να καλωσορίσω τον πρόεδρο της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας, τον κύριο Μάριο Ντράγκη. Σας ευχαριστούμε για την παρουσία σας σε αυτόν τον τρίτο νομισματικό διάλογο του έτους. Από τον τελευταίο νομισματικό διάλογο τον Μάιο η οικονομική διεύρυνση στην Ευρωζώνη έχει αποκτήσει μια θετική δυναμική και οι τελευταίες προβλέψεις δείχνουν ότι υπάρχει μια θετική επιτάχυνση της ανάπτυξης και γνωρίζουμε ότι πρέπει επίσης να εκτιμήσουμε βεβαίως στο πλαίσιο αυτό τις εξαιρετικές ε, επιδόσεις της ε, Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας στην οποία οφείλεται η καλύτερη κατάσταση στην οποία βρισκόμαστε σε μεγάλο βαθμό. Από την άλλη υπάρχει χαμηλή δυναμική όσον αφορά τον πληθωρισμό και αυτό είναι ε, ενδιαφέρον γιατί είναι και ένα ζήτημα ιδεολογικού χαρακτήρα, διανοητικού χαρακτήρα για το πώς ε, ε συνδυάζεται αυτή, αυτός ο χαμηλός πληθωρισμός όχι μόνο στην Ευρώπη με τις δυναμικές γύρω από την ανάπτυξη. Γνωρίζετε ότι στην τελευταία συνεδρίαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας του Σεπτεμβρίου αποφασίστηκε να παραμείνουν αμετάβλητα τα επιτόκια και να συνεχιστεί το πρόγραμμα αγορά στοιχείων του ενεργητικού έως το τέλος του 2017, ίσως και παραπάνω, αν κριθεί αναγκαίο. Και έως ότου το Δυτικό Συμβούλιο ε, δει ότι, πλέον, ότι υπάρχει πλέον μια ε, διαδρομή για την επίτευξη των στόχων όσον αφορά τον πληθωρισμό. Έχουν υπάρξει πολλές συζητήσεις βεβαίως όπως γνωρίζουμε όλοι αλλά δεν έχει ακόμα ε, συζητηθεί συγκεκριμένα ούτε το μέγεθος ούτε η διάρκεια του προγράμματος. Ξέρουμε ότι η συζήτηση αυτή θα γίνει κάποια στιγμή μέσα στο φθινόπωρο χωρίς να έχει ανακοινωθεί συγκεκριμένη ημερομηνία. Άρα ε, περιμένουμε ε, να γίνει αυτή η συζήτηση όπου θα υπάρξει και ένας ε, απολογισμός των προοπτικών, των οικονομικών προοπτικών αυτή τη στιγμή. Επίσης, έχουμε ζητήσει να συζητήσουμε με τον κύριο Ντράγκη δύο ακόμη στοιχεία. Το πρόβλημα της ενιαίας νομισματικής πολιτικής και της εφαρμογής της, καθώς και τις ε, προοπτικές του προγράμματος αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα. Είχαμε, κάνει, είχαμε προετοιμάσει και κάποια πολύ ενδιαφέροντα έγγραφα με σκοπό να υπάρξει μια συζήτηση όσον αφορά την αποκεντρωμένη εφαρμογή ή εκτέλεση αν θέλετε, άσκηση της νομισματικής πολιτικής, καθώς και το ζήτημα ορισμένων στοιχείων, πλευρών αυτής της πολιτικής, που υλοποιούνται, που ασκούνται σε, σε αποκεντρωμένη βάση. Αναφέρομαι συγκεκριμένα στον ELA. Άρα θα έχουμε την ευκαιρία να συζητήσουμε αν ε, προκρίνεται ή συζητείται ενδεχομένως ε, στο πλαίσιο αυτό μια πιο κεντρική διαχείριση των θεμάτων αυτών. Ε, ο πρόεδρος ε, Ντράγκη ε, μας έχει ενημερώσει ότι το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα βρίσκεται ήδη σε εφαρμογή. Έχουν υπάρξει κλήσεις για μεγαλύτερη διαφάνεια και βελτιώσεις στον τομέα αυτό της διαφάνειας και από την δική μας επιτροπή και με χαρά έχουμε διαπιστώσει ότι πράγματι έχουν σημειωθεί βήματα. Βεβαίως μπορούμε να συζητήσουμε και περαιτέρω ε, ε βήματα, χωρίς ωστόσο να πληγεί ο ε, καθ' αυτόν χαρακτήρας αυτού του ε, μέσου. Σας ευχαριστούμε λοιπόν για την παρουσία σας κύριε Ντράγκη. Έχετε το λόγο. Thank you, Mr. Ευχαριστώ, Πρόεδρε αξιότιμα μέλη τη Επιτροπή Οικονομικών και Ενωσιατικών Θεμάτων, κύριε και κύριοι. Χαίρομαι πολύ που ξανάρχομαι εδώ στην Επιτροπή σας ε, για την τρίτη ακρόαση του 2017. Πριν από ένα χρόνο συζητούσαμε από κοινού ε, την, ε, το μέτριο ρυθμό ανάκαμψης στην ζώνη του ευρώ και βλέπαμε μια μικρή μείωση της ορμής που, είχαμε κατόπιν του ε, δημοψηφίσματος του ε, τα τους τελευταίους 12 μήνες όμως η ανάκαμψη έχει επιταχυνθεί και διευρυνθεί και στηρίζεται από την αποτελεσματικότητα της νομισματικής μας πολιτικής. Στις σημερινές μου παρατηρήσεις θα μιλήσω για την σημερινή κατάσταση οικονομίας και το πώς την επηρεάζουν τα μέτρα νομισματικής πολιτικής που λαμβάνουμε. Η Επιτροπή σας μου ζήτησε να εστιάσω κυρίως σε δύο θέματα που σχετίζονται με τη νομισματική πολιτική της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Πιο συγκεκριμένα το πρόγραμμα αγοράς ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα, το CSPP, και την ε, εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής στην ζώνη του ευρώ. Η οικονομική μεγέθηση είναι πλέον σταθερή και ευρεία σε όλη την ζώνη του ευρώ, σε όλες τις χώρες του ευρώ και σε όλους τους τομείς. Η πραγματική ανάπτυξη, αύξηση του ΑΕΠ ήταν υψηλότερη από ό,τι περιμέναμε το πρώτο εξάμεινο του 2017 στο 2,3% ετησίως το δεύτερο τρίμηνο του έτους. Η οικονομία της ζώνης του ευρώ ε, επί 17 συνεχή τρίμηνα παρουσιάζει ανάπτυξη και οι τελευταίες πληροφορίες αναφέρουν ότι αυτό θα συνεχιστεί και στο προβλέψιμο μέλλον. Η ανάκαμψη αυτή ε, βασίζεται κυρίως σε παράγοντες σχετικούς με την εσωτερική αγορά, ενώ η αγορά εργασίας έχει βελτιωθεί σημαντικά. Η ανεργία έχει πέσει στα χαμηλότερα επίπεδα των τελευταίων 8 ετών. Ο αριθμός των εργαζόμενων στην ζώνη του ευρώ αυξήθηκε κατά περίπου σχεδόν 7 εκατομμύρια από τα μέσα του 2013. Αυτή η αύξηση των θέσεων εργασίας μαζί με την αύξηση του πλούτου των νοικοκυριών ε, στηρίζουν την ιδιωτική κατανάλωση, κατανάλωση στον ιδιωτικό τομέα. Επιπλέον βελτιώνεται και οι επενδύσεις ε, στηριζόμενες από τις πολύ ευνοϊκές ε, ε, ε συνθήκες που αφορούν τη χρηματοδότηση. Ε, οι, όλοι αυτοί οι παράγοντε μα καθιστούν πιο ισχυρού έναντι εξωτερικών παραγόντων. Σύμφωνα με τι δικέ μα οικονομικέ προβλέψει του Σεπτεμβρίου, η οικονομική μεγέθυνση θα συνεχίσει ε, άνω του δυνητικού προϊόντο σε ό,τι αφορά το μέλλον, μέλλον. Ε, το ετήσιο ΑΕΠ προβλέπεται ότι θα αυξηθεί κατά 2,2% το 2017, 1,8% το 2018 και 1,7% το 2019. Οι κίνδυνοι που σχετίζονται με την ε, ανάπτυξη στη ζώνη του ευρώ είναι ισορροπημένοι. Ταυτόχρονα αρνητικοί κίνδυνοι εξακολουθούν να υπάρχουν, κυρίως σχετίζονται με ε, παράγοντες στην παγκόσμια οικονομία, στις παγκόσμιες εξελίξεις και σε ξένες ε, χρηματαγορές η ανάπτυξη, η οικονομική ανάκαμψη πρέπει να βασιστεί ακόμα περισσότερο στην ε, ε, δυναμική του πληθωρισμού. Όπως έλεγα και παλιότερα, έχει εξαφανιστεί πλέον ο κίνδυνος του αποπληθωρισμού. Όμως, ε, μέτρα για την, για την αύξηση του πληθωρισμού δεν έχουν δώσει ακριβώς το επιθυμητό αποτέλεσμα. Ο συνολικός πληθωρισμός που ήταν 1,5% τον Αύγουστο αναμένεται ότι θα μειωθεί λίγο προσωρινά προς το τέλος του χρόνου, κυρίως εξαιτίας των εξελίξεων στον τομέα της ενέργειας. Αργότερα αναμένουμε ότι θα αυξηθεί και πάλι ο πληθωρισμός σταδιακά και θα φτάσει το 1,5% το 2019 σύμφωνα με τις προβλέψεις του προσωπικού της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Συνολικά, Όλο και περισσότερο είμαστε, γινόμαστε σίγουροι ότι ο πληθωρισμός τελικά θα φτάσει στα επίπεδα που έχουμε ως στόχο. Γνωρίζουμε όμως επίσης ότι ένα σημαντικό βαθμό νομισματικής ε, ε, χαλάρωσης είναι εξακολουθεί να, χρειάζεται προκειμένου να αυξηθεί ο πληθωρισμός στο επίπεδο που χρειάζεται. Επιπλέον βλέπουμε και κάποιες αβεβαιότητες σε ό,τι αφορά τον μεσοπρόθεσμο πληθωρισμό. Ε, κυρίως η πρόσφατη μεταβλητότητα στην ισοτιμία του ευρώ είναι ένας παράγοντας αβεβαιότητας που απαιτεί την στενή μας παρακολούθηση ε, προκειμένου να αξιολογήσουμε τις συνέπειες, τους, τις συνέπειες της μεταβλητότητας στον μεσοπρόθεσμο πληθωρισμό. Θα πρέπει λοιπόν να είμαστε ε, επίμονοι και υπομονετικοί η αύξηση του πληθωρισμού, μια ε, πάγια αύξηση του πληθωρισμού ε, που θα αυτοσυντηρείται απαιτεί ενίσχυση της οικονομίας συνολικά. Ε, και προφανώς χρειάζεται μια, ένας μεγάλος βαθμός νομισματικής χαλάρωσης ακόμα. Ε, γι' αυτόν τον λόγο φέτος, αργότερα, ε, το 2017, θα ξαναδιαρθρώσουμε τα όργανα που έχουμε έτσι ώστε ε, η, να στηρίξουμε την οικονομία της ζώνης του ευρώ και να ολοκληρώσουμε την μετάβαση σε μια καινούρια πορεία ισορροπημένης ανάπτυξης. Να σας πω δύο λόγια τώρα για το πρόγραμμα αγοράς πλουσιακών στοιχείων του εταιρικού εταιριών. Ε, η νομισματική πολιτική, τα μέτρα νομισματικής πολιτικής, τα οποία εφαρμόζουμε σταδιακά από τον Ιούνιο του 2014, ε, διευκόλυναν ε, σημαντικά την χρηματοδότηση ε, αυτό που είναι σαφές σήμερα και πολύ δύσκολο κανεί μπορεί να το αρνηθεί είναι ότι αυτή η νομισματική πολιτική οδηγεί όλο και περισσότερο σε ισχυρότερη οικονομική δραστηριότητα, ψηλότερα εισοδήματα και καλύτερες συνθήκε συνθήκες ε, απασχόλησης για τον πληθυσμό στη ζώνη του ευρώ. Ένα βασικό παραγόντας ήταν ε, η δυνατότητά μα ε, να ενεργοποιήσουμε μέτρα με συμβατικά μέτρα τα οποία έδωσαν πρόσθετη όθηση στον παραγωγικό τομέα. Για παράδειγμα, ε, η χρήση του τραπεζικού συστήματος, ε, η οποία μας βοήθησε πάρα πολύ ε, μέσω για παράδειγμα του προγράμματος EPP, δηλαδή προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων και ένα κομμάτι του οποίου είναι αυτό στο οποίο θέλω να εστιάσω που είναι το πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων ε, ε, ε, εταιριών. μαζί με τους τίτλους που προέρχονται από τιτλοποίηση και τις καλυμμένες ομολογίες, το ECSPP αποτελεί ένα σημαντικό συστοιχείο του προγράμματος αγοράς περιουσιακών στοιχείων. Μειώνοντας το κόστος χρηματοδότησης των μη ε, τραπεζικών εταιριών ε, κάνουμε πιο αποτελεσματική νομισματική μας πολιτική. Μέσω του CSPP το ευρωσύστημα από τον Ιούνιο 2016 έχει αγοράσει ομόλογα ε, ενός ε, μεγά, φάσματος ε, μη τραπεζικών εταιριών στη ζώνη του ευρώ που περιλαμβάνουν μεγάλες αλλά και μερικές μικρότερες εταιρείες. Μέχρι τώρα περίπου 110 δισεκατομμύρια ευρώ εταιρικών ομολόγων έχουν αγοραστεί από 200 περίπου εκδότες σε 20 χώρες, σε όλους τους τομείς ε, οικονομικής δραστηριότητας. Αυτές οι πληροφορίες βρίσκονται στο ίντερνετ, στο site της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας και στις δημοσίευσεις μας και ενημερώνονται τακτικά. Εξακολουθούμε να αναλύουμε δυνατότητες να μοιραστούμε ακόμα περισσότερες πληροφορίες με το κοινό ε, όσο αυτό μπορεί να βελτιώσει τη διαφάνεια χωρίς να υποσκάψει την αποτελεσματικότητα της νομισματικής μας πολιτικής. Χάρη στο πρόγραμμα αγοράς εταιρικών ομολόγων, εταιρείες στη ζώνη του ευρώ ε, είδαμε ότι βελτιώθηκε, βελτιώθηκαν πάρα πολύ οι δυνατότητε χρηματοδότηση που είχαν ε, όταν εκ, εκ, ε, κατά την έκθεση των ομολόγων του. Όμω, αυτέ οι βελτιώσεις που προέρχονται από το CSPP δεν περιορίζονται μόνο στις εταιρείε των οποίων τα ε, εταιρικά ομόλογα αγοράσαμε. επηρεάζουν και άλλες εταιρείε σε άλλους τομείς. Για παράδειγμα, τα σπρέ των αποδόσεων ε, των καλυμμένων εταιρικών ομολόγων που ε, δεν ε, αγοράζουμε, γιατί για παράδειγμα εκδίδονται από χρηματοοικονομικά ιδρύματα, έπεσαν αυτά τα spread σχεδόν 70 βαθμούς βάσης από το 1,25% το Μάρτιο 2016 στο 0,57% τώρα. Και αυτό από τότε που ανακοινώθηκε το πρόγραμμα CSPP. Τα spread των ε, εταιρικών ομολόγων ε, μη επενδυτικού βαθμού, που επίσης δεν είναι ε, δικαιούχοι επιλέξιμα, έπεσαν επίσης 262 πόντους βάσης, από το 5,59% το Μάρτιο του 2016 στο 2,97% σήμερα. Αυτές οι αγορές, ε, ε, προκειμένου αυτές οι αγορές να ενισχύσουν τη δραστηριότητα και τον πληθωρισμό, αυτές ε, πρέπει οι βελτιώσεις των χρηματοοικονομικών αγορών να περάσουν στις συνθήκες χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας, τους όρους χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας. Υπ' αυτή την έννοια έχουμε δει μια τέτοια μετάβαση σε βελτίωση των όρων χρηματοδότησης μικρών και μικρομεσαίων επιχειρήσεων. Όσο, περισσό, όσο όλο και περισσότερες εταιρείες αναζητούν ε, χρηματοδότηση από τις αγορές ε, οι εταιρείε ε, αποκτούν μεγαλύτερη δυνατότητα να δίδουν δάνεια σε μικρότερες εταιρείε που έχουν περισσότερο περιορισμένες δυνατότητες πρόσβασης σε πηγέ χρηματοδότηση. Συνεπώ, ο δανεισμός με μικρά, με χαμηλά με, ο δανεισμός από τράπεζες έχει πέσει, ε, τα επιτόκια δανεισμού από τράπεζες έχουν πέσει κατά 50 πόντους ε, βάσης από τότε που ανακοινώσαμε το CSPP. Ε, στην τελευταία μας έκθεση βλέπουμε ότι μικρότερες εταιρείε αντιμετωπίζουν καλύτερους, καλύτερες συνθήκες χρηματοδότησης και καλύτερη πρόσβαση. Το CSPP λοιπόν έχει ενισχύσει την αποτελεσματικότητα των αγορών περιουσιακών στοιχείων στην στις όρους χρηματοδότησης της πραγματικής οικονομίας και έχει ε, ευνοήσει τις θετικές εξέλιξεις πληθωρισμών. πληθωρισμό. Η υποστήριξη που προσφέρουν τα μέτρα μας, τα μέτρα πολιτικής, με όλα τα στοιχεία από την αγορά ε, τίτλων, στις συνθήκες της χρηματοδότησης, ως εκ είναι προφανής σε όλους τους τομείς και σε όλες τις χώρες της ζώνης του ευρώ. Με άλλα λόγια, βλέπουμε μια ομαλή μετάβαση, μετάδοση μάλλον, της πολιτικής μας, της ενιαίας νομισματικής πολιτικής. Ένα ενιαίο νόμισμα σημαίνει και ενιαία νομισματική πολιτική και έξι, έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο ε, λαμβάνει αποφάσεις για την επίτευξη του πρωταρχικού στόχου της διαφύλαξης της σταθερότητας των τιμών για την Ευρωζώνη στο σύνολό τη και επίσης θεσπίζει τις απαραίτητες κατευθυντήριες γραμμές για την εφαρμογή αυτών των στόχων. Ταυτόχρονα και σύμφωνα με το καταστατικό της, η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα προσφεύγει και στις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες στο βαθμό που θεωρείται απαραίτητος και σκόπιμος για την υλοποίηση των ε, δραστηριοτήτων που αποτελούν μέρος των καθηκόντων του ευρωσυστήματος. Οι εθνικές λοιπόν κεντρικές τράπεζες έχουν καθήκον να ακολουθούν τις κατευθυντήριες γραμμές και τις οδηγίες της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Αυτή η αποκεντρωμένη προσέγγιση λαμβάνει υπόψη την χρηματοοικονομική δομή της Ευρωζώνης, δηλαδή μια νομισματική ένωση που απαρτίζεται από κατακαιρματισμένες εθνικές χρηματοπιστωτικές αγορές. Και έτσι σε ένα τέτοιο περιβάλλον η στενή συνεργασία των Εθνικών Κεντρικών Τραπεζών με τις τράπεζες υπό, την, ε, υπό τον έλεγχό τους, στη δικαιοδοσία τους, φέρνει ωφέλη για την υλοποίηση της νομισματικής πολιτικής. Οι παραδείγματα μπορούμε να συλλέγουμε ακριβείς πληροφορίες από ευρύ φάσμα των εθνικών ε, ε, κεντρικών τραπεζών, εναρμονισμένα και προσαρμοσμένα στην ε, διάθεση πληροφοριών και την υλοποίηση της πολιτικής ε, του ε, Διοικητικού Συμβουλίου. Επιπλέον, οι Εθνικέ Κεντρικέ Τράπεζε γνωρίζουν καλά ποιες είναι οι ιδιαιτερότητε των επιχειρήσεων στην δικαιοδοσία τους και έτσι μπορούν να διαχειρίζονται τα στοιχεία ενεργητικού και τον τρόπο με τον οποίο θα πρέπει να χρησιμοποιούνται. Έτσι λοιπόν έχουμε μια αποκεντρωμένη ε, διαχείριση πολύ πιο αποτελεσματική από μια κεντρική προσέγγιση. Αφού δεν υπάρχει ενιαία, πραγματικά ενιαία αγορά κεφαλαίων, ε, ακόμη οι αγορές των ομολόγων εξαρτώνται σε μεγάλο βαθμό από τις ιδιαιτερότητες της κάθε εθνικής δικαιοδοσίας και από τις προτιμήσεις τους. Ε, μια επιτυχημένη βέβαια ένωση κεφαλαίων αγορών θα πρέπει να καταργήσει τις ε, ε, διακρίσεις μεταξύ του, τις διαχωριστικές γραμμές μεταξύ των δικαιοδοσιών με θετικά αποτελέσματα στον τρόπο υλοποίησης της νομισματικής μας πολιτικής και εν τέλει δεν πρέπει να λησμονούμε και τη βασική αιτία της ύπαρξης αυτής της νομισματικής ένωσης ήταν ακριβώς μια πιο ολοκληρωμένη ε, αγορά κεφαλαιακή και η εξασφάλιση των ωφελών ε, από για τις συνθήκες χρηματοδότησης σε όλη την Ευρωζώνη. Για να ολοκληρώσω λοιπόν, θα ήθελα να αναφερθώ στην αποκέντρωση και ιδιαίτερα να πω ότι οι μη τυποποιημένε ε, πολιτικές και τα μέτρα, τα μη τυποποιημένα που έχουμε εισαγάγει έχουν φέρει πολύ θετικά αποτελέσματα για τις εταιρείε αλλά και τα νοικοκυριά σε όλη την Ευρωζώνη. Ωστόσο δεν πρέπει να λησμονούμε τα προβλήματα και την κατάσταση που αντιμετωπίσαμε κατά το ε, χειρότερο σημείο της κρίσης, παραδείγματι θεσμικές αδυναμίες, οι διαρθρωτικές αδυναμίες ή υπορβολική ανάληψη κινδύνων συνέβαλαν σε, ένα αρνητικό, σε μια αρνητική εικόνα ε, στροβιλιζόμενη μεταξύ των ε, κεντρικών τραπεζών και των ε, τραπεζών σε διάφορες χώρες. Και αυτό οδήγησε σε κίνδυνο και για τη σταθερότητα των τιμών στην Ευρωζώνη που ήταν ο βασικός στόχος που θέλαμε να εξυπηρετήσουμε. Έτσι λοιπόν πρέπει να κλείσει αυτός ο φαύλος κύκλος τώρα. Έχουμε πάρει αντίστροφες, ε, έχουμε στοιχεία για αντίστροφες τάσεις με θετική, ε, θετικό αντίκτυπο σε όλες τις χώρες, καταγραφόμενο. Ε, όλοι έχουν ωφεληθεί από αυτά τα μέτρα που υποστηρίζουν την ανάπτυξη όλη την Ευρωζώνη και έτσι εξασφαλίζουν ένα πεδίο για υγιή επάνωδο του πληθωρισμού σε επίπεδα σύμφωνα με τους στόχους μας. Ωστόσο, παρότι υπάρχει αυτή η κυκλική προσαρμογή και προχωρεί, έχουμε ακόμη διαρθρωτικά ζητήματα που θα πρέπει να αντιμετωπίσουμε. Ε, τα επόμενα χρόνια, λοιπόν, υψηλότερο επίπεδο ε, διαρκούς και συνεπούς σύγκλησης αλλά και ενισχυμένης ανθεκτικότητας θα είναι απαραίτητο για να επιτευχθεί μια καλύτερη, καλύτερα λειτουργούσα οικονομική νομισματική ένωση και αυτό σημαίνει από τη μία πλευρά ότι θα λαμβάνονται αποφάσεις πολιτικής από τις εθνικές κυβερνήσεις που το στόχο θα έχουν την ε, απεμπλοκή του παραγωγικού δυναμικού των οικονομιών μας και από την άλλη πλευρά θα πρέπει να ληφθούν και αποφασιστικά μέτρα για την ε, διακυβέρνηση Οικονομικής και Σωματικής Ένωσης που θα είναι σύμφωνα με τους στόχους μας. Ευχαριστώ πολύ για την προσοχή σας. Ο Πρόεδρος, ευχαριστώ πολύ κύριε Ντράγκη. Πολύ ενδιαφέρουσα η παρουσίαση. Και βεβαίως αναμένουμε αυτά τα περαιτέρω αποφασιστικά μέτρα ώστε το σύστημα διακυβέρνησης της Ευρωζώνης να εξυπηρετεί πλήρως τους στόχους του. Ταυτόχρονα η υπομονή και η επιμονή που εκφράζεται ως κατευθυντήρια αρχή με στόχο και τον επαναπροσδιορισμό αλλά και ένα ευρύ επίπεδο ε, νομισματικής προσαρμογής μας οδηγεί στην ολοκλήρωση της, κεφαλαϊκής, της Ένωσης Κεφαλαϊκών Αγορών και βλέπουμε ότι μπορεί να έχει και θετικό αντίκτυπο σε ε, επιχειρήσεις οι οποίες δεν εντάσσονται στους όρους της αγοράς ομολόγων. Μπορούμε να περάσουμε τώρα στις ερωτήσεις-απαντήσεις. Ο κύριος Χέις είναι ο πρώτος ομιλητής. Κύριε Ντράγκη, σας ευχαριστώ για την παρουσία σας. Δύο ερωτήματα έχω. Το ένα αφορά τον στόχο πληθωρισμού που έχετε θέσει εδώ και έχει αρκετό καιρό και ένα δεύτερο ε, ε ζήτημα που αφορά την ποσοτική χαλάρωση. Για το πρώτο θέμα. Είπατε πρόσφατα ότι οι προβλέψεις για τον πληθωρισμό της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας έχουν αναθεωρηθεί προς τα κάτω για το 2018 και 2019 λόγω της ισχύω του ευρώ έναντι του ντάρ, του δολαρίου. Βλέπουμε ότι υπάρχει μία ε, ανωδική πορεία του ευρώ έναντι του δολαρίου και αυτό λόγω των ε, δυσκολιών που αντιμετωπίζει η Αμερικανική ε, οικονομία. Αυτά τα δύο στοιχεία, ισχυρό ευρώ, αδύναμη ή, εν πάση περιπτώσει, προβλήματα στην Αμερικανική οικονομία, θεωρείτε ότι είναι επιτεύξιμος ο στόχος του 2%? αν πράγματι επιμένετε σε αυτόν. Μετά, για το ζήτημα του, του, ε, του, 33% στο πρόγραμμα προσωπικής χαλάρωσης, η ΕΚΤ κατέχει ακόμη ε, μεγάλο ε, τμήμα των ομολόγων. Στην Ιρλανδία, στην Πορτογαλία, στη Γερμανία υπάρχει, βρισκόμαστε κοντά σε αυτό το όριο του 33%. Αλλά το ερώτημα μου είναι πώς αυτές οι χώρες μπορούν να μην πληγούν δυσανάλογα από αυτό το όριο των 33%, του, του 33%. Ε, με βάση τις, ε, τις αγορές της, ε, της ΕΚΤ. Μήπως έχετε εξετάσει πιθανή αύξηση αυτού του ορίου σε περίπτωση, για παράδειγμα, πώλησης των ομολόγων σε μια χώρα μήπως ε, ε, θα, θα μπορούσαμε με μια τέτοια κίνηση να ανακόψουμε τυχόν αρνητικές εξελίξεις, ιδίως για τις χώρες που είναι πολύ κοντά στο, όριο. Ευχαριστώ. Πράγματι, αναθεωρήσαμε προς τα κάτω. Και τώρα προβλέπουμε ε, ότι αυτή η διαδρομή του πληθωρισμού θα κάνει ένα μικρό νι. Ε, θα κατέβει, μετά θα ξανανεύει λίγο. Αυτό ε, οφείλεται κυρίως ε, στις τιμές του πετρελαίου. Κάτι στο οποίο ε, η, αναβάθμιση και η ενίσχυση του ευρώ, ανατίμηση του ευρώ το τελευταίο, το τελευταίο διάστημα έχει βεβαίως συμβάλει. Επίσης, έχω πει ότι η συνταγματική ισοτιμία δεν είναι ε, στόχος πολιτικής. Είναι απλά ένα στοιχείο που λαμβάνουμε υπόψη στο πλαίσιο της ανάπτυξης και της μεγένθησης δεν είναι εύκολο να προσδιορίσει κανείς ε, ποια είναι η, η ε, ε, επιρροή της ανατίμησης αυτής στην, στο προβλεπόμενο ποσοστό του, του πληθωρισμού. Υπάρχουν τρεις παράγοντες τουλάχιστον. Πρώτον είναι η αδιαμφισβήτητη ανάκαμψη που παρατηρείται στην Ευρωζώνη. Και εδώ υπάρχει, υπάρχει μια ε, γενική τάση ε, ε, που αντικατοπτρίζεται και στον πληθωρισμό. Υπάρχουν όμως και άλλοι δύο παράγοντες. Πρώτον, αναμένονται διαφορετικές οικονομικές και νομισματικές πολιτικές στις διαφορετικές δικαιοδοσίες. Και τρίτον, ε, τρίτος παράγοντας σχετίζεται με τη γενική βελτίωση του κλίματος που επικρατεί παγκόσμια ε, απέναντι στην Ευρωζώνη. Και αυτό οφείλεται εν μέρη και σε πολιτικούς λόγους, στις πολιτικές εξελίξεις των τελευταίων 6-7 μηνών και βλέπετε ότι ναι, η συναλλαγματική ισοτιμία πράγματι σε ένα βαθμό αντικατοπτρίζει και τις ε, πολιτικές εξελίξεις που έχουν υπάρξει το τελευταίο διάστημα στην Ευρωζώνη. Έτσι λοιπόν υπάρχει μια αύξηση της στην Ευρωζώνη. Είναι δύσκολο να καθορίσουμε και να ποσοτικοποιήσουμε ποιος από αυτούς τους τρεις παράγοντες έχει ε, επηρεάσει την σημερινή κατάσταση περισσότερο. Πάντως και οι τρεις παράγοντες ε, έχουν επηρεάσει την κατάσταση του πληθωρισμού και έτσι το Διοικητικό Συμβούλιο είπε ότι θα, παρακολουθεί, θα συνεχίσει να παρακολουθεί την, ε, την κατάσταση με μια κάποια ανησυχία. Όσον αφορά τα, τα ομόλογα, εμείς εξακολουθούμε να πιστεύουμε ότι ε, χάρη στην οικονομική πολιτική που εφαρμόζουμε θα επιτύχουμε τους στόχους μας και ε, η διαδρομή του πληθωρισμού θα ε, συνεχίσει να συγκλίνει με έναν βιώσιμο και συνεπή τρόπο. Αλλά θα πρέπει να είμαστε, να επιδείξουμε και υπομονή και επιμονή όσον αφορά την υλοποίηση της, της ε, νομισματικής μας πολιτικής. Για το δεύτερο ερώτημα, πράγματι ε, μετρούμε όλα τα ομόλογα που έχουμε στο χαρτοφυλάκιο μας αυτών των κρατών μελών ε, που αναφέρατε στο ε, όριο του 33%. Όχι, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει συζητήσει πιθανή αλλαγή αυτού του όριου. Για να απαντήσω στο ερώτημα σας. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ η κυρία Περέζ. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ε, μετά από ερώτηση επιτροπή μας ε, ε, σε ό,τι αφορά τον αποκεντρωμένο χαρακτήρα τη εφαρμής τη νομισματική πολιτικής είπατε κάποια πράγματα. Η Κομισιόν πριν από λίγες μέρες δημοσίευσε μια σημαντική πρόταση αναθεώρησης της λειτουργίας της παρακολούθησης επιτήρησης των τραπεζών δεν φαντάζομαι ότι έχετε παρακολουθήσει από κοντά ε, την λειτουργία των ε, υπηρεσιών ε, της Ευρωπαϊκής Ένωσης πώς μπορούν αυτές οι υπηρεσίες, αυτοί οι οργανισμοί της Ευρωπαϊκής Ένωσης να ευθυγραμμιστούν περισσότερο με τη δράση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ε, προφανώς δεν είστε ο, ο κατεξοχήν υπεύθυνο για αυτά τι υπηρεσίε, αλλά ίσω μπορείτε να απαντήσετε. Ε, εγώ είμαι επίση μία από τους ευρωβουλευτέ που υπέγραψαν την επιστολή που σας ε, ζητούσε περισσότερη διαφάνεια στο, ε, στη λειτουργία του προγράμματος CSPP. Ε, εσείς ο ίδιος είπατε ότι η πρόθεσή σας είναι να βελτιωθεί η διαφάνεια. Ε, προφανώς δεν έχουμε κανένα σκοπό να ε, θέσουμε υπό αμφισβήτηση το πρόγραμμα της ποσοτικής χαλάρωσης, αλλά αντιθέτως να το ενισχύσουμε θέλουμε. Ε, είπατε ότι μελετάτε, εξετάζετε την δυνατότητα να αυξήσετε τη διαφάνεια, δηλαδή να, κάνετε, να δημοσιεύσετε περισσότερα στοιχεία. Μπορείτε να μας πείτε δύο λόγια παραπάνω για αυτές τις προθέσεις. Ε, καλωσορίζουμε το, την έκθεση ε, αυτή, την πρόταση αυτή της Κομισιόν που περιλαμβάνει αλλαγές στην ε, λειτουργία της Ευρωπαϊκής Αρχής ε, Επιτήρησης. Το νέο πλαίσιο. Έχει κάνει το συνολικό σύστημα πιο αποτελεσματικό, πιο ανθεκτικό και εμείς ε, που καθορίζουμε την νομισματική πολιτική ευνοούμαστε από αυτό. Γιατί με τον τρόπο αυτό έχουμε μεγαλύτερη σιγουριά, ε, ε, πιο μακροπρόθεσμα από ότι θα είχαμε αν το τραπεζικό σύστημα ήταν λιγότερο ασφαλές. Οπότε στηρίζουμε αυτή την την πρόταση της ε, Κομισιόν. Ε, σε ό,τι αφορά την ε, δική μας λειτουργία δεν βλέπουμε να μας επηρεάζει. Ε, αλλά θέλουμε οι προτάσεις Κομισιόν να ε, είναι πραγματικά χρήσιμες και γι' αυτό το λόγο οποιασδήποτε προτάσεις ε, γίνουν για να βελτιώσουμε τη λειτουργία μας είναι καλοδεχούμενες. Well, we want to discuss... Ένα από τα θέματα που έχουμε συζητήσει είναι να δώσουμε πιο σημαντικό ρόλο στην Διευθύνουσα Επιτροπή, το, τη Steering Committee. Το ε, SRB ε, είναι μια ε, συμβουλευτική επιτροπή. Έχει ως στόχο να εκδίδει γνωμοδοτήσεις και να χτυπάει καμπανάκια, να μας προειδοποιεί. Ε, αυτό θέλουμε να ε, διατηρήσουμε. Ε, το άλλο, η άλλη που μπορεί να της δοθεί είναι να είναι ένας, μια επιτροπή όπου η, όλα τα μέλη της επιτροπής, Διευθύνουσας Επιτροπής να μπορούν να ανταλλάσσουν απόψεις και γνώμες για το πώς μπορούν να βελτιωθούν τα πράγματα. Και αυτό μπορεί να γίνει από την ESRB. Το έχει, έχει προταθεί ήδη. Ε, μιλάμε για συντονισμό, έτσι, όχι για λήψη αποφάσεων. Να είναι ένα χώρο στον οποίο να γίνεται ανταλλαγή απόψεων. Επίσης θα πρέπει να προβλέψουμε για την ολοκλήρωση της ε, τραπεζικής αγοράς, ε, την οποία των ε, κεφαλαιογορών, ε, όλα αυτά θα συζητηθούν εκεί, θα μπορούν να συζητώνται. Σε ό,τι αφορά τη διαφάνεια, ε, νομίζω ότι είμαστε διαφανείς. Και έχουμε, κάνει, και έχουμε βελτιώσει την κατάσταση ε, από τον Ιούνιο δεν έχουμε τίποτα εναντίον της ε, αποκάλυψης πληροφοριών υπό την προϋπόθεση ότι αυτό, αυτή η δημοσίευση, αυτή η δημοσιότητα ε, δεν θα παρεμποδίζει την εφαρμογή της νομισματικής μας πολιτικής. Ε, δεν θέλουμε μέσω αυτής της αποκάλυψης και της δημοσιότητας οι αγορές να κινούνται εναντίον μας. Σας είπα εταιρείε, ε, πάνω από χίλια εταιρικά ομόλογα. Ε, δεν θέλουμε ε, να δείξουμε ότι προτιμούμε την α ή β εταιρεία, το α ή β ομόλογο. Οπότε τώρα σε ό,τι αφορά αυτό που ζητήθηκε να κατονομάζουμε συγκεκριμένους εκδότες. Πιστεύω ότι αυτό ε, και θα δυσκόλευε το δικό μας έργο, αλλά και θα δημιουργούσε προβλήματα μεταξύ των εταιρεών, γιατί η μία θα πληροφορεί το για, τις, ε, για τη χρηματοδότηση της άλλης. Όμως, υπό την προπόθεση ότι τα μέτρα μας είναι αποτελεσματικά, θα προχωρήσουμε προς την αύξηση της διαφάνειας. Ευχαριστώ. Thank you, Chairman. Welcome, Mr. Ευχαριστώ Πρόεδρε και καλώς ήρθατε κύριε Ντράκη. Θα αρχίσουμε εδώ να συζητούμε την ετήσια έκθεση της ΕΚΤ σύντομα και μάλιστα εγώ είμαι εισηγητής εκ μέρους του Κοινοβουλίου. Θέλω λοιπόν ε, να διατυπώσω κάποιες ερωτήσεις και να ρωτήσω ποια είναι η γνώμη σας για κάποιες ιδέες που κυκλοφορούν σε σχέση με τη διαφάνεια κυρίως. Καταρχά, κυκλοφορεί μια πρόταση για την αποτροπή συγκρούσεων συμφερόντων που λέει ότι θα πρέπει να δημοσιεύει ε, δηλώσεις οικονομικών συμφερόντων για τα μέλη του Διοικητικού της Συμβουλίου, η ΕΚΤ. Και ότι επίσης η Επιτροπή Δεοντολογίας δεν θα πρέπει πλέον να τίθεται υπό την Προεδρία του πρώην Προέδρου της ΕΚΤ. Θα ήθελα λοιπόν να μου πείτε ποια είναι η γνώμη σας για τα δύο αυτά θέματα. Απάντηση. Ε, ευχαριστώ και βεβαίω μα απασχολούν και τα δύο αυτά θέματα. Καταρχήν δεν έχουμε αντίρρηση ούτε για την ούτε για την άλλη πρόταση, αλλά βεβαίω θα πρέπει να τα συζητήσουμε με του συναδέλφου στο Διοικητικό Συμβούλιο. Κοιτάξτε, έχω ετοιμάσει μια ακόμη ερώτηση για την Κίνα, γιατί ήταν, η απάντηση μου δώσαν αυτή ακριβώ περίμενα. Έχουμε λοιπόν την έκθεση BITS που λέει ότι υπάρχουν κάποιες ανησυχίες σε σχέση με ε, άνευ προηγουμένου ποσοστά ε, επιτοκίων χρηματοδότησης χρέους ε, για την Κίνα. Πώς βλέπετε λοιπόν εκεί την οικονομική κατάσταση και τι μπορεί να φέρει μια ευνίδια επιβράδυνση της οικονομίας της Κίνας για τις δικές μας ευρωπαϊκές οικονομίες. Μπορεί αυτό να οδηγήσει μια παγκόσμια κρίση δηλαδή και βλέπετε κάποιο κίνδυνο σχετικά πιθανό ή πόσο πιθανό. Απάντηση. Ναι. Είδαμε την έκθεση της BIS και έχουμε δει βέβαια και τις δικές μας μελέτες για την Κίνα, δύο είναι τα στοιχεία. Καταρχάς η παγκόσμια ε, οικονομική σταθερότητα και δεύτερον οι συνέπειες για τις οικονομίες της Ευρωζώνης, για την οικονομία της Ευρωζώνης. Πρώτον, εμείς θεωρούμε ότι οι οικονομικές αρχές της Κίνας είναι σε θέση με επάρκεια να αντιμετωπίσουν και έχουν ήδη αρχίσει να αντιδρούν σε κάθε επίπεδο και μέτωπο που έχει εντοπίσει η ΒΑΙΑ στις αναλύσεις της. Ως προς τις συνέπειες. Και σημειώνω ότι δεν πρόκειται για έναν ε, μακρινό κίνδυνο. Είχαμε ήδη ε, στην αρχή της διαδικασίας 2015 την έκφραση φόβων για σοβαρή επιβράδυνση της κινέζικης οικονομίας. Ωστόσο τώρα έχουμε πολύ διαφορετικές συνθήκες. Για το 2015, και αυτό ήταν ένας από τους λόγους για τους οποίους χρειάστηκε να ενισχύσουμε το πρόγραμμα νομισματικής πολιτικής μας. Τώρα λοιπόν έχουν αλλάξει συνθήκες σημαντικά. Η οικονομική ανάκαμψη, συνεχιζόμενη οικονομική ανάπτυξη ε, στηρίζεται κατά βάση και κατά κύριο λόγο σε εγχώριες πηγές, εγχώρια κατανάλωση και εγχώριες επενδύσεις, όπου βεβαίως τα χαμηλά επιτόκια συμβάλλουν. Το πραγματικό διαθέσιμο εισόδημα ενισχύεται λόγω της ενισχυμένης απασχόλησης. Και έτσι η επιβράδυνση ή μια δυσμενής εξέλιξη στις παγκόσμιες οικονομικές συνθήκες ασφαλώς δεν θα κριθεί θετική, αλλά πάντοτε θα έχει τόσο σοβαρές επιπτώσεις όσο θα μπορούσε να έχει πριν από δύο χρόνια. Ευχαριστώ. Κύριος Γουαλτιέρη, συνεχίζετε αν θέλετε. Χαίρομαι που κρίνετε θετικά τις δράσεις των κινέζικων αρχών, ε, των οικονομικών αρχών. Στα όσα τεκταίνονται στη Βόρεια Κορέα, για να μιλήσουμε για την παγκόσμια οικονομία. Εκεί που μιλούσαμε για οικονομικά μπαζούκα, τώρα μιλούμε για άνθρωπο πύραυλο. Πώς το βλέπετε αυτό, κύριο Δράγκη. Όταν ε, λέμε, ολοκληρώνοντα τη συνεδρίασή μα τις συνεδριάσεις μας, ότι η εξωτερική ζήτηση υποστηρίζει ακόμη την ε, οικονομία της Ευρωζώνης, αλλά υπάρχει κίνδυνος ε, αρνητικός, αυτός ο κίνδυνος ο αρνητικός είναι βασικά γεωπολιτικού χαρακτήρα. Γκουαλτιέρη. Ωρα Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Σας καλωσορίζω και πάλι εδώ στην Επιτροπή και εγώ θα ήθελα να σας ρωτήσω, να σας θέσω δύο ερωτήματα. πέραν της συνήθους ε, νομισματικής πολιτικής, για τα κρυπτονομίσματα. Είναι πολύ καυτό ζήτημα. Η Κίνα έχει απαγορεύσει την έκδοση και την ε, ε, συναλλαγή ε, με τέτοια νομίσματα. Αντίστοιχα το Μεξικό εκδίδει νομοθεσία προκειμένου να ρυθμίζονται οι εταιρείες fintech και ο αντιπρόεδρος της ΕΚΤ είπε ότι Πρόκειται για ένα ε, εργαλείο ε, κερδοσκοπίας και μάλιστα συνέκρινα αυτά τα νέου είδους νομίσματα, τα ψηφιακά, ε, με, την, με τις, με τις τουλίπες πριν από κάποιους αιώνες στην Ολλανδία. Τι πιστεύετε ότι πρέπει να γίνει, ποια είναι τα βήματα που θέλετε να κάνετε. Ε, τίνεται περισσότερο στο, ε, στην κινέζικη πλευρά, στην κινέζικη στάση που θέλει να τα απαγορεύσει ή ε, συμφωνείτε πιο πολύ με τους Ιάπωνες που θέλουν να ρυθμιστεί αυτό το ζήτημα. Επίσης, για τις κατευθυντήριες γραμμές για ε, τα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα FinTech. σύμφωνα με αυτές τις κατευθυντήριες γραμμές, αυτού του είδους εταιρείε πρέπει να πληρούν υψηλότερα κριτήρια ε, κεφαλαιακής επάρκειας σε σχέση με τα παραδοσιακά τροπο, ε, ε, τραπεζικά ιδρύματα. Αυτό αποτελεί μειονέκτημα για τις, ε, για τις ευρωπαϊκές εταιρείες που δραστηριοποιούνται σε αυτόν τον τομέα. Και επίσης πώς ε, γίνεται αυτό να συνάδει, ε, αυτός ο κανόνας, αυτοί οι κατευθυντήριες γραμμές να συνάδουν με την αρχή οι ίδιοι κανόνες για ίδιες υπηρεσίες. Ενδεχομένως ε, θα μπορούσε να, αποτελεί, να, να πει κανείς ότι πρόκειται για ε, μειονεκτική μεταχείριση αυτών των εταιριών. Για το πρώτο ερώτημα, απάντηση. Πρέπει να ε, ρωτήσουμε είναι, είναι, ποιοι είναι οι υλικοί κίνδυνοι που θέτουν αυτά τα bitcoin στην ε, πραγματική οικονομία. Πρώτον, μέγεθος, ε, αποδεκτότητα από, τον, από τους χρήστες και αντίκτυπος των bitcoin στην πραγματική οικονομία. Αν εξετάσουμε και τους τρεις διάβλους, θα δείτε ότι πράγματι είναι πρόημο να θεωρήσουμε ότι πρόκειται για μέσο πληρωμής, το μέσο πληρωμής του μέλλοντος. Πρέπει να το δούμε σε μεγαλύτερο βάθος. Ε, με ρωτήσατε τι έχει αποφασίσει η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα. Δεν έχουμε κάνει τέτοια συζήτηση, ούτε έχουμε αρμοδιότητα να ρυθμίσουμε αυτό το ζήτημα, νομοθετικά προφανώς. ούτε έχουμε κάνει κάποια θεσμική συζήτηση για το θέμα αυτό. Υπάρχουν διάφορε απόψεις που έχουν εκφραστεί, Εσεί αναφερθήκατε σε μία από αυτέ. Πιο γενικά, και αυτό ε, απαντά και στο δεύτερο ερώτημά σας, είναι το εξής. Η βασική μα μας ανησυχία ε, με όλες αυτές τις καινοτομίες ε, στον ε, τομέα των χρηματοπιστωτικών, όχι μόνο τα bitcoin αλλά και άλλα, είναι ε, ο έθρος χαρακτήρας όσον αφορά τους ε, κυβερνοκινδύνους. Και εκεί επικεντρώνουμε τη δουλειά μας. Και αυτό βεβαίως ισχύει σε όλων των ειδών της καινοτομίας. Με ρωτήσατε γιατί οι κεφαλαιακές απαιτήσει ε, στις κατευθύνες γραμμές για τις εταιρείες FinTech είναι υψηλότερες από ότι για άλλα χρηματοπιστωτικά ιδρύματα. Συμφωνώ απολύτω μαζί σα. Οι ίδιοι κανόνε, οι ίδιε υπηρεσίε, οι ίδιε απαιτήσει. Με την προπόθεση ότι βεβαίω είναι οι ίδιοι και οι κίνδυνοι. Και σύμφωνα με τι κατευθείαν γραμμέ τη ΕΚΤ, εκτιμούμε ότι οι κίνδυνοι δεν είναι πάντοτε οι ίδιοι. Αλλά συμφωνώ μαζί σας ότι πρέπει να το εξετάσουμε σε μεγαλύτερο βάθος το θέμα αυτό. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, πρόεδρε, λέει ο κ. Κάρθη. Στην επισκέψη στην Ιρλανδία πολύ πρόσφατα, την πρώτη από όταν έγινε γίνατε πρόεδρος της ΕΚΤ, ορισμένες από τις παρατηρήσεις σας σχετιζόντουσαν ε, με τις φούσκες ακίνησης περιουσίας. Είπατε ότι η ΕΚΤ δεν έχει εντοπίσει τέτοιου είδους φούσκες στην Ευρωζώνη, καινούριες φούσκες στην Ευρωζώνη στο σύνολό της γιατί δεν, έχουν αυξηθεί, έχουν αυξηθεί πολύ τα δάνεια, τα στεγαστικά δάνεια. Ε, ε, υπάρχουν όμως ε, κάποιες ενδείξεις σε συγκεκριμένα κράτη-μέλη και ιδιαίτερα στην Ιρλανδία. Ε, υπάρχει έλλειψη προσφοράς, ιδιαίτερα σε κοινωνική στέγη, ε, κάτι που έχει οδηγήσει σε σημαντική αύξηση των τιμών πάνω από 12% σύμφωνα με τον ΟΣΑ φέτος. Ε, επίσης έχει αυξη, έχουν αυξηθεί πολύ οι χορηγήσεις ε, το 2017. Η ΕΚΤ βλέπει αυτές τις ενδείξεις και έχετε άποψη για το τι χρειάζεται προκειμένου να αποφύγουμε μια καινούρια τέτοια φούσκα. Και αν έχω χρόνο να ρωτήσω και το εξή ό,τι αφορά τον επιχειρηματικό τομέα και το πρόγραμμα αγοράς ε, εταιρικών ομολόγων και τη σχέση αυτού του προγράμματος με τις μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Γνωρίζω ότι πολύ συχνά λέτε ότι το πρόγραμμα αυτό είναι θετικό επειδή αγοράζοντα εταιρικά ομόλογα μεγάλων εταιριών ε, η ΕΚΤ ε, διευκολύνει τις τράπεζες ε, να δανείζουν χρήματα σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις. Μπορείτε όμως να το ποσοτικοποιήσετε αυτό. Μπορείτε να μας αποδείξετε με στοιχεία ότι συμβαίνει πράγματι αυτό. Ότι δηλαδή τα χρήματα τα οποία χρησιμοποιούμε την αγορά εταιρικών ομολόγων φτάνουν και στην πραγματική οικονομία και, όχι, και δεν είναι ένας απλός μηχανισμός να ευνοούμε τις μεγάλες επιχειρήσεις. Ευχαριστώ. Thank you. Κύριος σε ό,τι αφορά την ενδεχόμενη ύπαρξη φούσκας των, στον τομέα της, ε, των ακινήτων, θα πρέπει να κάνουμε διάκριση ανάμεσα στα συστημικά φαινόμενα και τα τοπικά φαινόμενα. Σε ορισμένες χώρες πράγματι, και μάλιστα σε ορισμένες πόλεις θα έλεγα, βλέπουμε ότι οι τιμές των ακινήτων αυξάνονται. Και συχνά αυτές οι αυξήσεις σχετίζονται, ξεκινούν από πολύ χαμηλά επίπεδα. Μερικές φορές βλέπουμε αυξήσεις από νορμάλα, από κανονικά επίπεδα, αλλά πολλές φορές είναι από πολύ χαμηλά, υποτιμημένα επίπεδα. Το φαινόμενο αυτό περιορίζεται σε συγκεκριμένες πόλεις και συγκεκριμένες χώρες. Δεν είναι συστημικό ζήτημα. Δεν έχει γενικευθεί. Πλην όμως μιλήσουμε και για φούσκες, θα πρέπει να σκεφτούμε μήπως αυτή η αύξηση τιμών της εκείνης περιουσίας ε, συνοδεύεται και από ε, εξίσου ανησυχητική αύξηση των στεγαστικών δανείων. Δηλαδή, η μόχλευση. Η μόχλευση αυξάνεται, γιατί αυτό ήταν ένα χαρακτηριστικό της οικονομίας πριν, της κρίση, πριν την κρίση και δεν περιοριζόταν μόνο στην, στα ακίνητα. Το, δεν βλέπουμε όμως αυτή την αύξηση. Τα στεγαστικά δάνεια αυτή τη στιγμή εξακολουθούν να είναι αρκετά χαμηλά. Αυξάνονται βέβαια σταδιακά, αλλά το συνολικό ποσό είναι πολύ πολύ χαμηλότερο από αυτό που είχαν πριν την κρίση. Και ταυτόχρονα η πραγματική οικονομία εξακολουθεί να χρηματοδοτείται έτσι ώστε να αναπτύσσεται. Οπότε δεν εντοπίζουμε κάποιο συστημικό κίνδυνο. Δεύτερον, πολύ συχνά ο λόγος αυτών των αυξήσεων στις τιμές των ακινήτων έχει σχέση με ελλείψεις στη μειωμένη προσφορά. Για παράδειγμα, μειωμένη προσφορά ε, κοινωνικών ε, κατοικιών. Ε, αν οι αυξήσει των τιμών ε, αρχίσουν να μας ανησυχούν, τι θα κάνουμε, θα αλλάξουμε την νομισματική μας πολιτική. Η απάντηση είναι όχι, σαφέστατα όχι, γιατί δεν πρόκειται για συστημικό ζήτημα. Ε, αυτό που μας ενδιαφέρει μας είναι η συστημική κίνδυνη. Η, ε, η Κεντρική Τράπεζα της Ιρλανδίας από το 2015 έχει ένα σύστημα προληπτικής εποπτείας και το αναθεώρησε και το 2016. Και άλλες χώρες έχουν, διαθέτουν παρόμοια, παρόμοια συστήματα προληπτικής εποπτείας. Για παράδειγμα, οι 100 Η Γαλλία το σκέφτεται. Και άλλες χώρες. Οπότε νομίζω ότι με αυτόν τον τρόπο θα πρέπει να αντιδράσουμε σε ε, τοπικές υπερτιμήσεις. Μπορεί, αν ψάξουμε, να εντοπίσουμε υπερβολές, αλλά στο σύνολο της Ευρωζώνης η στέγη δεν δείχνει να είναι υπερτιμημένη τουλάχιστον όχι σε ό,τι αφορά τις οικογένειε. Τώρα, μπορεί για εμπορικά κίνητα να έχουμε τέτοια φαινόμενα. Η ESRB, η Επιτροπή, ε, Ευρωπαϊκή Επιτροπή Συστημικού Κινδύνου, ε, πριν από ένα χρόνο ε, έστειλε μια προειδοποίηση, αν θυμάμαι καλά, σε οκτώ χώρες για, για το θέμα της υπερβολικής υπερτίμησης επαγγελματικών ακινήτων. Τώρα, Πολλές φορές έχουμε αναρωτηθεί και μάλιστα στην αρχή του προγράμματος αγοράς εταιρικών ομολόγων αν αυτό θα βελτίωνε τις ε, πιστοτικές, τους πιστοτικούς όρους ε, χρηματοδότησης των μικρομεσαίων επιχειρήσεων, ε, επιχειρήσεων εξίσου με ε, αυτή των μεγάλων επιχειρήσεων. Και αυτό που διαπιστώσαμε είναι ότι η βελτίωση ήταν ε, ε, πάρα πολύ σημαντική, όχι μόνο για τις μεσαίες επιχείρησεις, αλλά και για τις μικρομεσαίες. Ε, ακόμα και για αυτές τις επιχειρήσεις που εκδίδουν ομόλογα, αλλά που δεν είναι επιλέξιμα για το πρόγραμμα μας, το ε, CSPP. Δηλαδή και εταιρείε των οποίων τα ομόλογα δεν αγοράζουμε, είδαν ότι τα spread των ομολόγων τους μειώθηκαν πολύ. Τώρα, εταιρείε οι οποίες ε, απευθύνονται σε ζητούν τραπεζικό δανεισμό και δεν εκδίδουν ε, ομόλογα στις κεφαλαίες αγορές και αυτές ευνοήθηκαν. Δεν είναι εύκολο βέβαια να το ποσοτικοποιήσουμε, αλλά το καλύτερο μέτρο, ο καλύτερος δείκτης ποσοτικοποίησης και αυτού του προγράμματος και των άλλων ε, μέτρων μας είναι ε, οι, ε, οι χορηγήσεις των τραπεζών. Οι χορηγήσεις των τραπεζών ε, ή μάλλον τα επιτόκια των χορηγήσεων των τραπεζών σε μικρομεσαίες επιχειρήσεις έχουν μειωθεί πολύ σε όλη την Ευρωζώνη, ανεξάρτητα αν ε, αγοράζουμε πολλά εταιρικά ομόλογα της συγκεκριμένη χώρας ή όχι. τα επιτόκια μειώθηκαν, χορηγήσεων μειώθηκαν και στην Ισπανία πολύ και στην Ιταλία και αλλού. Δεν ισχυρίζομαι ότι αυτό αντικατοπτρίζει μόνο τα αποτελέσματα του προγράμματος αγοράς εταιρικών ομολόγων. Υπάρχουν και άλλοι παράγοντες. Thank you. Uh, Scott Cato. Ευχαριστώ κύριε Σκοτ Κέιτο. Πρόεδρε ευχαριστώ. Σε προηγούμενους γύρους του νομισματικού διαλόγου σας είχα επισημάνει το θέμα των ε, ε, απολεσθέντων πόρων, ε, στοιχείων ενεργητικού και θέλαμε να ακούσουμε ποια ήταν η προσέγγισή σας και βεβαίως σε σχέση και με, τις, με τους κλιματικούς κινδύνους. Έχετε λοιπόν πει ότι θα δώσετε για τα μία αξιοποιήσιμα στοιχεία ενεργητικού απαντήσεις γραπτές, ε, περιμένουμε να δούμε ρόλο, ε, απάντηση και σε σχέση με τις κλιματικές αλλαγές, γιατί στο άρθρο 2 των συμφωνιών αναφέρεστε και στην διαφύλαξη διατήρηση σε επίπεδο μέχρι δύο βαθμούς υψηλότερο από την περίοδο πριν από τη βιομηχανική ε, των, ε, της θερμοκρασίας και συγκράτηση των αερίων θερμοκηπίου, των όγκων αερίων θερμοκηπίου. Μπορείτε λοιπόν να μας πείτε αν συνεχίζετε να αγοράζετε από επιχειρήσεις, ομόλογα επιχειρήσεις οι οποίες όμως έχουν συμφέροντα στην εξαγωγή, εξόριξη και εκμετάλλευση ορυκτών ε, πόρων και καυσίμων και αν απελευθερωθούν τέτοιου είδους στοιχεία ε, μπορείτε να μας βεβαιώσετε ότι δεν πρόκειται να, να τα επανεπενδύσετε σε ε, επιχειρήσεις που εκμεταλλεύονται ρηκτούς πόρους. Επίσης μπορεί να υπάρξει κάποια ε, μετάβαση σε επενδύσεις σε πράσινη οικονομία. Μπορώ να πω ότι προβλέπω ήδη την απάντηση ότι είναι πολιτικές οι και τα λοιπά και μπορώ να το δεχτώ. Ένας οικονομολόγος όμως θα σας έλεγε ότι πρόκειται για οικονομικές στρεβλώσεις, λαμβανέτε αποφάσει δηλαδή ανάλογα με, ε, που σχετικές με τα ομόλογα που θα αγοράσετε. Αυτή τη στιγμή όμως ασκείται με τι επιλογέ αυτές και πολιτική. Επιλέγετε δηλαδή που θα πάνε τα, ε, που θα πάει ρευστότητα. Άρα υπάρχει επίδραση, πολιτικός ρόλος και στις δραστηριότητες της τράπεζας και αυτό το οποίο μας απασχολεί εδώ και σε αυτόν τον έλεγχο είναι αν είναι επαρκές αυτό ή αν θα πρέπει να υπάρχει μεγαλύτερη υποχρέωση λογοδοσίας για τις αποφάσεις που λαμβάνει η Κεντρική Τράπεζα. Απάντηση. Ευχαριστώ. Ας μην λησμονούμε λοιπόν ότι έχουμε μία εντολή που είναι η σταθερότητα των τιμών και αυτήν εξυπηρετούμε. Πέραν όμως του πρωταρχικού αυτού στόχου της σταθερότητας των τιμών, η ΕΚΤ υποστηρίζει τις γενικές πολιτικές και τους στόχους Ευρωπαϊκής Ένωσης, μεταξύ των οποίων το άρθρο 3 της συνθήκης συμπεριλαμβάνει την αηφόρο ανάπτυξη της Ευρώπης με στόχο υψηλό επίπεδο προστασίας και βελτίωσης της ποιότητας του περιβάλλοντος. Ως εκ τούτου η ΕΚΤ αναγνωρίζει και εντοπίζει τις προκλήσεις της κλιματικής αλλαγής και τη σημασία των πολιτικών που στόχο έχουν να την αντιμετωπίσουν. Και άρα, ναι, υποστηρίζουμε τις αποφάσεις που λαμβάνονται σε, σε διεθνή ή σε ευρωπαϊκά κέντρα αποφάσεων οι πολιτικές αυτές πρέπει να ενσωματώνονται στα μέτρα και το υφιστάμενο βέβαια και με βάση βέβαια το εφιστάμενο ρυθμιστικό πλαίσιο. Κάθε πιθανή αλλαγή στο ρυθμιστικό πλαίσιο ή την προληπτική ε, νομοθεσία για την αντιμετώπιση κλιματικής αλλαγής θα πρέπει να είναι και αιτιολογημένη προληπτικά και να υποστηρίζουν τον πρωταρχικό στόχο. Ευχαριστώ να επανέλθω, αν μου επιτρέπετε κυρία Σκοτκάτο, ε, στην αρχική μου ερώτηση, γιατί μίλησατε για την εντολή σας. Επαρκεί αυτή η εντολή όταν λαμβάνονται αποφάσεις για το πρόγραμμα αγοράς τίτλων και άλλες μορφές ε, χαλάρωσης, ε, ποσοτικής χαλάρωσης ε, σε σχέση με τις προτεραιότητες για τις ε, ροές ρευστότητα σε όλη την Ήπειρο. Δηλαδή η πολιτική, εμείς που είμαστε εδώ, Έχουμε επαρκή δυνατότητα επίδραση στον τρόπο με τον οποίο λαμβάνονται οι αποφάσεις σα. Απάντηση. Κοιτάξτε, αυτό που κάνουμε όταν σχεδιάζουμε τα κριτήρια επιλεξιμότητας για το πρόγραμμα τίτλων, αγορά τίτλων, ήταν το εξή. Τα σχεδιάσαμε κατά τρόπο αρκετά ευρύ, ώστε να μπορούμε και να αγοράζουμε τίτλου σαν αυτού του οποίου σα αναφέρεστε. Αυτό προσπαθούμε να κάνουμε. Αυτό κάνουμε. Και έτσι όπως είπα μόλις τώρα, υποστηρίζουμε αυτόν τον τρόπο και σεβόμαστε το άρθρο 3 της συνθήκης που αναφέρεται ρητά στην αηφορία και την ποιότητα του περιβάλλοντος. Ας μην ξεχνούμε. Δηλαδή, καταρχήν, συμφωνούμε απόλυτος μαζί σας. Αλλά έχουμε σαν πρώτη και κύρια την εντολή μας, την εντολή της νομισματικής, της ε, συγγνώμη, σταθερότητας των τιμών. Ε, και βεβαίως υπάρχουν πολιτικές αποφάσεις τις οποίες εμείς δεν επηρεάζουμε και δεν είναι δικής μας αρμοδιότητας. Σας ευχαριστώ. Κύριος Βάλλη. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ τον Μάριο Ντράγκη για το χρόνο που μας αφιερώνει. Μια ερώτηση λοιπόν για το tapering το οποίο προεξαγγέλλεται ή τέλος πάντων μέχρι το 2018 θα έχει προχωρήσει η ΕΚΤ πώς σκοπεύει αυτό το μέτρο της ελάφρυνσης της ε, αγοράς τίτλων να το υποστηρίξει, να το εξασφαλίσει και οι αποδόσεις στις περιφερειακές χώρες πώς σκοπεύει να αποτρέψει να γίνουν υπερβολικά βαρύς βαριές οι αποδόσεις για τους εθνικούς προϋπολογισμούς έτσι ώστε να μην συνεχιστούν τα μέτρα λιτότητας τα οποία στόχο έχουν να ε, μειώσουν το spread και τα επιτόκια για τους ε, τίτλους. Και δεύτερον, ένα σχόλιο, μου επιτρέπετε, για τις εκλογές στη Γερμανία. Θα σας ρωτήσω λοιπόν να μου πείτε, θεωρείτε ότι μπορεί αυτό να επιταχύνει μία ε, έξοδο από το πρόγραμμα αγοράς τίτλων. Κύριο Στράκη. Ευχαριστώ πολύ. Για το δεύτερο δεν μπορώ πραγματικά να σας απαντήσω. Θα ήταν προώρο και βέβαια εκτός των αρμοδιοτήτων μας το να κάνουμε κάποιο σχόλιο για τις εκλογές στη Γερμανία. Δεν μπορώ να κάνω. Είναι εκτός εντολής μου να κάνω σχόλια για τις εκλογές στις διάφορες χώρες. Για το πρώτο ερώτημα. Πρώτα απ' όλα το Συμβούλιο δεν έχει λάβει, το Διοικητικό Συμβούλιο δεν έχει λάβει απόφαση καμία απόφαση. Είπαμε ότι πρόκειται να συζητήσουμε την πολιτική μας, ε, πολιτική μας την νομισματική, τις επιλογές μας νομισματικής πολιτικής για το μέλλον. Είπα πάντως ότι στην επόμενη συνεδρία του Οκτωβρίου θα έχουμε προσδιορίσει τις αδρές γραμμές αυτής της πολιτικής. Για κάποια ζητήματα όμως πρέπει να πω ότι θα ήταν πρόωρο να ρωτήσει κανείς τι είδους συνέπειες μπορεί να φέρουν στα Ιταλικά εντωμεταξύ ή τα επιτόκια των ε, ομολόγων. Ωστόσο πρέπει να λαμβάνουμε υπόψη ότι η εντολή, η πρωταρχική εντολή της ΕΚΤ είναι η σταθερότητα των τιμών σε όλη την Ευρωζώνη. Και κυρίω πρέπει να κοιτάξουμε το κατά πόσο ο πληθωρισμό συγκλίνει κατά τρόπο βιώσιμο και ανεξάρτητο προς ένα επίπεδο κοντά στο 2% ή χαμηλότερο το 2%. Επαναλαμβάνω στα Ιταλικά, Εντολή μας είναι η διαφύλαξη της σταθερότητας των τιμών με ένα πληθωρισμό έως και κοντά στο 2%, ο οποίος πληθωρισμός θα μπορεί να είναι αυτοσυντηρήτος, χωρίς δηλαδή τη δική μας νομισματική υποστήριξη. Το ίδιο ισχύει για τις χώρες της περιφερειακής της Ευρώπης που όμως δεν είναι ο κύριος στόχος μας. Ο κύριος στόχος μας, κύριο καθήκον και εντολή μας είναι η σταθερότητα των τιμών και πάνω σε αυτό εστιάζονται οι στόχοι μας. Ε, δεύτερη ερώτηση από τον κύριο Βάλλη. Ο πληθωρισμός όμως αυξάνεται. Και έτσι μήπως ε, σκέφτεστε ότι θα μπορούσατε να προχωρήσετε σε ελάφρυνση των μέτρων αγοράς των ομολόγων και μήπως δεν συνεχιστούν τα μέτρα αυτά και για το 2018 ή για μακρύτερη περίοδο. Κύριος Δράκη. Με ρωτάτε τι θα απαντήσουμε στο επόμενο Διοικητικό Συμβούλιο. Όπως είπα, είναι προώρο να μου κάνετε τις ερωτήσεις. Αφήστε μας να συζητήσουμε μεταξύ μας και στην επόμενη ακρόαση της Επιτροπής σας να σας δώσω απαντήσεις. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μπερνάρ Μονό έχει το λόγο. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Ε, οι συνθήκες ορίζουν ότι το ευρώ ε, έχει κλείσει να μετατραπεί σε νόμισμα όλων των ευρωπαϊκών κρατών μελών και των κρατών που σκοπεύουν να ενταχθούν στην Ένωση, πλην της αυτοεξαιρούμενης Δανίας βεβαίως, ε, μετά τις ε, δηλώσεις του κυρίου Μοσκοβισή στην ε, ομιλία για την κατάσταση Ένωση πριν από δύο εβδομάδες, ο κύριος Γιουνκέρ ξεκάθαρα είπε ότι αποσκοπεί η Ένωση και η Επιτροπή στην εξασφάλιση της συμμετοχής στο ευρώ με ενδεχόμενη ακόμα και την δυνατότητα προενταξιακού μέσου διευκόλυνση δηλαδή τεχνικής προς την ένταξη κάποια χώρα στη ζώνη, στη ζώνη του ευρώ. Δηλαδή μου φαίνεται ότι πάλι κάνουμε τα πράγματα ανάποδα. Είναι μεγάλε ε, οι προκλήσει μακροοικονομικέ. Η υιοθέτηση της, ε, του ενιαίου νομίσματο, από ό,τι μα λέει και η μακροοικονομία μπορεί να γίνει μόνο όταν έχουν πραγματικά συγκλίνει οι οικονομίε, Οικονομίε οι οποίε πράγματι δεν είχαν συγκλίνει στην, κατά την εισαγωγή του ευρώ του 1999 και που αποδεικνύεται πως έχουν φέρει ακόμα μεγαλύτερε αποκλήσει και διαφορέ μεταξύ των κρατών ε, της Ευρωζώνης με ιδιαίτερο και χαρακτηριστικό παράδειγμα το ε, υπερβολικό πλεόνασμα της Γερμανίας. Όταν λοιπόν ε, αποφασίσουν τα κράτη για μια αμετάκλητη ισοτιμία του νομίσματός τους με την γερμανική οικονομία, μήπως δημιουργούν ακόμα μεγαλύτερες αποκλήσεις και ε, διαφορές ε, μεταξύ των κρατών, της Ευρω... των κρατών και οικονομιών της Ευρωζώνης που οδηγούσαν σε ακόμα μεγαλύτερη αποσταθεροποίηση. Μήπως θα έπρεπε να αποφύγουμε την βεβαιασμένη ε, ένταξη στο ενιαίο νόμισμα. Μήπως θα έπρεπε να κοιτάμε περισσότερο και ως μόνη προτεραιότητα την οικονομική σύγκληση. Εάν λοιπόν ε, αυτός είναι ο στόχος, ο δεύτερος, θα έπρεπε πιστεύετε να ορίζονται συγκεκριμένα χρονοδιαγράμματα για την ένταξη των κρατών στην Ευρωζώνη. Ορισμένα μάλιστα από αυτά, όπως η Πολωνία, η Τσεχική Δημοκρατία, η Ουγγαρία, η Σουηδία φαίνονται ικανοποιημένα από την διαφύλαξη, από την δυνατότητα διατήρησης των εθνικών ε, μοχλεύσεων στις ισοτιμίες τους. Μήπως λοιπόν θα έπρεπε να δείξουν μεγαλύτερη αποφασιστικότητα για την προσχώρηση αυτή στην ε, Ευρωζώνη τα κράτη αυτά. Ευχαριστώ για την απάντησή σας. Όχι, όχι βέβαια. Όπως είπατε, όλα τα κράτη-μέλη, με την, εξε... με την εξαίρεση της Δανίας βεβαίως και του Ηνωμένου Βασιλείου, πρέπει να προσχωρήσουν στην ε, ζώνη του ευρώ μόλις ε, εκπληρώσουν τις ε, οικονομικές και νομικές απαιτήσεις. Οι εθνικές κυβερνήσεις βεβαίως πρέπει να επιδείξουν και τη βούληση, την πολιτική για την προσχώρησή τους στην Ευρωζώνη. Δεδομένου αυτού, η προσχώρηση μιας χώρας στην ε, Ευρωζώνη αποφασίζεται από το Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης λαμβάνοντας υπόψη την αξιολόγηση της Κομισιόν και της ε- Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας όσον αφορά την εκπλήρωση αυτών των νομικών και οικονομικών απαιτήσεων. Και αυτή η αξιολόγηση βασίζεται αποκλειστικά στα κριτήρια σύγκλησης που κατοχυρώνονται σαφώς στο άρθρο 140 της Συνδίκης για τη Λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Η τελευταία αξιολόγηση της ΕΚΤ εκδόθηκε τον Ιούνιο του 2016 και βάσει αυτής της αξιολόγησης καμία χώρα δεν εκπληρούσε όλα τα κριτήρια που θεσπίζονται βάσει της συνθήκης. Και έτσι το Συμβούλιο δεν έλαβε σχετική απόφαση για την προσχώρηση χώρας ε, στην Ευρωζώνη. Άρα, η ΕΚΤ θα επανέλθει σε έλεγχο και εξέταση των κριτηρίων σύγκλησης, όπως αυτά κατοχυρώνονται στη συνθήκη, και θα επανέλθει με νέα έκθεσή της για αυτό το ζήτημα, την οποία και θα υποβάλει στο Συμβούλιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης και όλο αυτό βλέπετε να γίνει του χρόνου, το 2018. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Γιούνκερ έτσι κι αλλιώς δεν μίλησε ποτέ να, για εξαναγκασμό κάποιας χώρες, αλλά για υποστήριξη και πολιτική βούληση που πρέπει να εκφραστεί. Ο κύριος Λάγκεν, αν δέχεται να, ζητή, να πάρει τον, τη θέση του κύριος Λούκε, γιατί πρέπει να φύγει. Ευχαριστώ. Θα μιλήσω γερμανικά, λέει ο κύριος Λούκε. Κύριε Ντράγκη, το Συνταγματικό Δικαστήριο της Γερμανίας απέστειλε κατάλογο ερωτημάτων όσον αφορά το PSPP της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. και εκεί αναφέρεται ότι αυτό το PSPP αντίκειται στα άρθρα 119, 127 και στα άρθρα 17-24 του εσωτερικού κανονισμού του καταστατικού της Ευρωπαϊκής Τράπεζας, διότι τα, οι σορευτικοί όγκοι του PSPP γίνονται τόσο μεγάλοι έπειτα από κάποιο διάστημα που γίνεται, καθίσταται αυσύμβατη η κατάσταση με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Το, το ερώτημά μου είναι ε, το εξή. Εσείς πιστεύετε ότι υπάρχει κάποιο ορισμένο μέγιστο ε, όριο για το PSPP από το οποίο και έπειτα το PSPP αντίκειται στην Ευρωπαϊκή Νομοθεσία και αν πιστεύετε ότι υπάρχει ένας τέτοιος μέγιστος όγκος για το PSPP, θα ήθελα να μου πείτε πώς μπορεί κανείς να το προσδιορίσει αυτό το μέγιστο όγκο. Ποια κριτήρια δηλαδή χρησιμοποιεί η ΕΚΤ προκειμένου να προσδιορίσει, να προσδιορίσει αυτό το μέγιστο όγκο. Αν δε πιστεύετε ότι δεν υπάρχει τέτοιο μέγιστο όριο, ότι δηλαδή μπορεί απεριόριστα η ΕΚΤ να αγοράζει κρατικά ομόλογα, να μας το πείτε ξεκάθαρα, σας παρακαλώ. Ήταν ε, εύκολα δομημένη η ερώτησή μου, οπότε μπορείτε να ξεκινήσετε την απάντησή σας λέγοντας ναι ή όχι και στη συνέχεια να το αιτιολογήσετε. Ευχαριστώ. Η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ε, έχει σημειώσει την απόφαση του Συνταγματικού Δικαστηρίου και εμείς θεωρούμε ότι η διεύρυνση αυτού του προγράμματος αγοράς βρίσκεται εντύπτει εντό της ε, ε, αρμοδιότητές μας και δεν πρόκειται να προβούμε σε κανένα περαιτέρω σχόλιο. Το PSPP βρίσκεται σε πλήρη λειτουργία και εξέλιξη σύμφωνα με τις αποφάσεις που έχει λάβει το Διοικητικό Συμβούλιο της ΕΚΤ. Κύριε Πρόεδρε, δεν σας ζήτησα να σχολιάσετε την διαδικασία που βρίσκεται υπό εξέλιξη. Σας ζήτησα να ε, μου σχολιάσετε τη συμβατότητα του PSPP με την Ευρωπαϊκή Νομοθεσία. Γνωρίζετε ότι το PSPP έτσι όπως το έχετε ε, ε, διαμορφώσει, αν συνεχιστεί χωρίς κανένα περιορισμό, χρονικό ή άλλο, Ξέρετε πολύ καλά ότι ε, ε, ε, θέλω να μου απαντήσετε αν μια τέτοια συνέχιση απεριόριστη του, του συγκεκριμένου προγράμματο είναι συμβατή με το δίκαιο της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Το ε, πρόγραμμα αγορά του επιχειρηματικού τομέα, ομολόγων του επιχειρηματικού τομέα αποτελεί κατά τη γνώμη μας εμπίπτη στην αρμοδιότητά μας. Ναι. Άρα, λέει ο κ. Λούκε, πιστεύετε ότι δεν πρέπει να υπάρχουν περιορισμοί ως προς τους όγκους του PSPP. Μιλώ μόνο για αυτό και όχι για το πρόγραμμα αγοράς στοιχείων του ενεργητικού γενικά. Άρα η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα μπορεί απεριόριστα να συνεχίζει το συγκεκριμένο πρόγραμμα. Αυτό είπατε. Όχι, υπάρχουν όρια ως προς τις εκδόσεις και τους εκδότες. Αυτός είναι όμως ο μόνος περιορισμός αφορά τους εκδότες, δεν αφορά τον όγκο. Ρωτάει ο κύριος Λούκε. Είπα ότι υπάρχουν ζητήματα ως προς την έκδοση, υπάρχουν περιορισμοί ως προς την έκδοση και τους εκδότες. Κύριε, προσπαθείτε να μου βάλετε πράγματα στο στόμα για να βγείτε αύριο στα πρωτοσέλιδα των εφημερίδων. Ε, θέλω να μιλήσω γερμανικά, λέει ο κ. Λούκε. 25 δευτερόλεπτα έχετε. Είμαι βουλευτής και νομίζω ότι λογοδοτείτε σε εμάς για να... και σας ρωτώ αν υπάρχει όριο ως προς τον όγκο για το PSPP. Ξέρω ότι μου απαντήσατε για το, για το ε, για τους εκδότες. Μα γνωρίζετε, λέει ο κύριος Ντράγκη, ε, ποια είναι αυτά τα όρια που έχουν θεσπιστεί. Μπορείτε να τα υπολογίσετε και μόνος σας. Κύριε Λάγκεν, ευχαριστώ πολύ κύριε Πρόεδρε και εγώ θα μιλήσω γερμανικά. Θέλω να ε, ρωτήσω κάτι σχετικό με αυτό που είπε ο κύριος για το όριο του 33%. Είπατε ότι δεν έχει τεθεί ε, επιτάπητος ακόμα αυτό το θέμα. Συζητείτε όμως και κάτι που συνδέεται με αυτό που ρώτησε ο κύριος Λούκε. Πρόκειται για ε, σταθερό όριο ή μπορεί και να υπάρξει υπέρβαση αυτού. Δεύτερο ερώτημα. Ανάκαμψη, ανάπτυξη, δυναμική πληθωρισμού θετική, δεν, έχει αποσοβηθεί ο κίνδυνος από πληθωρισμού, ανατίμηση του ευρώ. Ε, Πότε πιστεύετε εσείς ότι θα είναι η κατάλληλη στιγμή για μια αλλαγή της νομισματικής πολιτικής και την αχαλάρωση. Και τρίτο ερώτημα. Έχουμε συζητήσει πολλές φορές και μάλιστα είχαμε συμφωνήσει ότι πρόκειται για πολιτική απόφαση. Το πώς θα μπορέσουν να βελτιωθούν οι συνθήκες ε, ο πρόεδρος ε, Γιούγκερ έχει κάνει κάποιες προτάσεις, ε, προϋπολογισμός του ευρώ, ενίσχυση αρμοδιοτήτων, Ευρωπαϊκό Νομισματικό Ταμείο, ευρώ για όλους. Το ερώτημά μου είναι, αυτός είναι κατά τη γνώμη σας ο σωστός δρόμος για, την, ε, για, για τις πολιτικές μεταρρυθμίσεις. Και τελευταίο ερώτημα. Είχατε ε, στις αρχές του χρόνου απαντήσαμε είναι και στον συνάδελφο Φέρμπερ ότι οι δύο μεγάλοι στόχοι ε, βασίστηκαν ε, στην ε, συνήθη την, την κανονική εξέλιξη και δεν πηγάζουν από τα προβλήματα που δημιούργησε η κρίση. Τι ακριβώς εννοείτε με αυτή την, την κανονική εξέλιξη. Μπορείτε να επαναλάβετε σας παρακαλώ λέει ο κύριος Δράκη, το, την... Οι στόχοι για, τον, για το Target 2 που αυξήθηκαν ε, πάνω από 700, 800 δισεκατομμύρια ευρώ. Ε, είχαν μειωθεί και τώρα έχουν αρχίσει να ξανανεβαίνουν. Είχατε απαντήσει ότι δεν ήταν τα διαρθρωτικά προβλήματα της οικονομικής κρίσης, αλλά ήταν ότι πρόκειται για μια φυσιολογική εξέλιξη ε, το γεγονός ότι βρίσκονται πάλι σε αν, ανωδική πορεία. Θέλω να μου εξηγήσετε αυτόν τον όρο που χρησιμοποιήσατε, φυσιολογική εξέλιξη. Για την πρώτη σας ερώτηση, έχουμε το 33% ως όριο. Δεν έχουμε ποτέ συζητήσει να το αλλάξουμε. Δεν έχω να σας αναφέρω τίποτα γι' αυτό. Για τη δεύτερη ερώτησή σας. Πότε θα αλλάξουμε... Ναι, ε, έχουμε κριτήρια. Ε, είναι ε, ο πληθωρισμός ε, θέλουμε να συγκλίνει με το στόχο μας ε, με τρόπο ε, ε, αυτοδιατηρούμενο α, και διαρκείας και για μεγάλο χρονικό διάστημα. δεν έχουμε φτάσει ως εκεί, έχουμε πει ότι ο πληθωρισμός θα μειωθεί και μετά θα ξαναυξηθεί σε ένα σχήμα V τα επόμενα χρόνια. αυτό το προφίλ εξαρτάται από αλλαγές στις τιμές του πετρελαίου. και σε αλλαγές στην ε, ισοτιμία, των νομισμό και Ε, αλλά αν εξαιρέσουμε την ενέργεια και τα, τρόφιμα, ε, θα δούμε ότι ο πληθωρισμός έχει αυξηθεί λιγάκι τους τελευταίους μήνες. Όμως αυτό δεν αποτελεί αποδεικτικό στοιχείο αύξησης, πραγματικής αύξησης. Ε, γιατί οι μισθοί δεν έχουν αυξηθεί επαρκώς, ε, αυξάνονται σε μέτριο ρυθμό και γι' αυτό το λόγο και ο πληθωρισμός δεν ακολουθεί. Ο στόχος πάντως είναι ο πληθωρισμός να συγκλίνει με το στόχο μας για μεγάλο χρονικό διάστημα και να αυτό συντηρείται. Τώρα, για τις εξελίξεις στο Target 2. Είναι αλήθεια ότι δεν αποτελούν αποτέλεσμα τέλεσμα των εξελίξεων κατά τη διάρκεια της, νομισματικής, της οικονομικής κρίσης. Πολλές από αυτές τις εξελίξεις, όχι όλες, πολλές από αυτές, οφείλονται στο ίδιο το πρόγραμμα ποσοτικής χαλάρωσης και αγοράς περιουσιακών στοιχείων ε, που εφαρμόστηκε μέσω της αγοράς ε, ομολόγων. Γι' αυτό το λόγο εν μέρη βλέπουμε υψηλότερες εξελίξεις στο Target 2 η βελτίωση της εμπιστοσύνης στη ζώνη του ευρώ και η βελτίωση των οικονομικών συνθήκων σε όλη την ζώνη του ευρώ που παρατηρείται αυτή τη στιγμή, αυτά τα δύο, αυτοί οι δύο παράγοντες θα μας ενισχύουν όλο και λιγότερο. υπάρχει όμως ένα θέμα ε, λειτουργίας του σύστηματος πληρωμών στην Ευρωπαϊκή Ένωση. Ευχαριστώ. Ο κ. Φερνάντεθ. καλώ ήρθατε κύριε Ντράκη. Ο κ. Λάγκεν. Ε, ε, ε, δεν προηγήθηκε μόνο του κ. Λούκε. Ο κ. Λούκε προ, μπήκε πριν από όλου εμάς. Ε, δεν έγινε μια ανταλλαγή σλότ. Ο κ. Λούκε απλώ προηγήθηκε όλων των υπολείπων. Αυτό ήθελα να πω. Τέλο πάντων, μετά από αυτό το σχολείο να πω το εξή. Ε, βλέποντας την αναθεώρηση των προβλέψεων για την εξέλιξη του πληθωρισμού, ε, ε, βλέπουμε και την εξέλιξη στην ισοτιμία του ευρώ. Ε, για δύο ακόμα χρόνια ε, φαίνεται ότι θα διατηρηθεί το πρόγραμμα. Περιμένουμε βέβαια τις ε, αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Τράπεζας. Βλέπουμε ότι υπάρχουν ε, πιέσεις ως προς την εφαρμογή της νομισματικής πολιτικής από την ΕΚΤ. Αλλά να σας ρωτήσω το εξής. Μίλησατε για την αποκέντρωση της νομισματικής πολιτικής. Να σας ρωτήσω ακριβώ για αυτό το πράγμα, για την ε, αποκεντρωμένη εφαρμογή του ELA, του Μηχανισμού ρευστότητα για τις Τράπεζε. Δημιουργεί η αποκέντρωση αυτή προβλήματα στην, στην τραπεζική ενοποίηση. Ο υποθετή τη Τράπεζα Ισπανία έλεγε αυτή τη βδομάδα ότι η Λαϊκή Τράπεζα έχει περιουσιακά στοιχεία επαρκή έτσι ώστε να εξακολουθήσει να διαθέτει πρόσβαση στον ELA. Και από ό,τι φαίνεται τα κριτήρια της ε, Τράπεζας της Ισπανίας είναι διαφορετικά από τα κριτήρια άλλων εθνικών κεντρικών τραπεζών σε ό,τι αφορά ε, την αποδοχή περιουσιακών στοιχείων ως εξασφαλίσεων προκειμένου να δοθεί την ΑΒ τράπεζα πρόσβαση στον ELA. Αυτή η διαφορά κριτηρίων μπορεί να επηρέασε ε, την, τον αποκλεισμό πρόσβαση της ε, Banco Popular στον ELA. Δηλαδή αν αυτή η συγκεκριμένη τράπεζα βρισκόταν σε μια άλλη χώρα που εφάρμοζε τον ELA με διαφορετικά κριτήρια θα μπορούσε η τράπεζα να εξακολουθήσει να είναι ζωντανή, να, να έχει πρόσβαση στον ELA. Ε, λαμβάνοντας το όσα είπατε ε, για την αποκέντρωση ε, της τη ε, της Επιτροπή, Επιτροπής μήπως θα πρέπει ταυτόχρονα αυτή η αποκέντρωση να γίνει με ενιοποίηση, ενοποίηση των κριτηρίων εφαρμογή του ELA στι διάφορε χώρες. Φύγεται ένα θέμα το οποίο έχει συζητηθεί επανειλημμένος ε, στην, στο Δυτικό Συμβούλιο. Θα ήταν ε, φυσιολογικό να θεωρήσουμε ότι έχοντας ε, μία ενιαία εποπτική αρχή και μία αρχή ε, ε, και ανάκτησης των τραπεζών να έχουμε και ένα ενιαίο ELA. Αλλά ο ELA είναι αποκεντρωμένος και οι αποφάσεις του και η εφαρμογή του βαραίνουν τις Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες. Η συμφωνία μεταξύ όλων των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου είναι ο η ΕΛΕΗ να μπορεί να χρησιμοποιηθεί όπως θέλει η Εθνική, ε, όπως θέλει Κεντρική Τράπεζα από την προϋπόθεση ότι αυτό δεν θα υποσκάπτει τις συνολικές, τις γενικότερες αρχές της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Ε, δεν έχουμε, το θέμα αυτό συζητήθηκε πριν από ένα χρόνο τελευταία φορά, αλλά δεν βλέπω να γίνεται κανένα είδου αλλαγή σε αυτό τον κανόνα τον, τον, το επόμενο χρονικό διάστημα. Η σημερινή εφαρμογή του ELA όμως είναι πρόβλημα στην ενοποίηση της, ε, ε, της Τραπεζικής Ένωσης στη δημιουργία της Τραπεζικής Ένωσης. Κάποια στιγμή στο μέλλον θα πρέπει να το εξετάσουμε, λέει ο κ. Δράγκη. Υπάρχουν κάποιοι οι οποίοι ε, το θεωρούν ως πρόβλημα, ειδικά μετά την ορία του SSM και τη Ευρωπαϊκής Επιτροπή Συστημικού Κινδύνου. Η Εθνική Κεντρική Τράπεζα συνήθως έχει όλες τις πληροφορίες, είναι πολύ πιο πληροφορημένη από την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα ή κάποια άλλα ε, κεντρικά όργανα. Γι' αυτό το λόγο οι Εθνικές Κεντρικές Τράπεζες ε, δυσκολεύονται να παραχωρήσουν αυτή την εθνική αρμοδιότητα. Θα ήταν όμως φυσιολογικό πράγματι να έχουμε ένα μόνο όργανο το οποίο θα λαμβάνει όλες τις αποφάσεις για τον ELA. Λογικό φαίνεται. Ο κ. Χόπμαν. Ευχαριστώ. Θα ήθελα να επανέλθω σε ερωτήσεις του κ. Λάγκεν. Το μικρόφωνο παρακαλούμε. Το μικρόφωνο είναι κλειστό. Ο κύριος Χόκμαρκ δεν ακούγεται. I was ecological here. Uh, a lot of things... Ναι, πολλά πράγματα στη ζωή δεν είναι τα ίδια ως, όπως πριν. Και το ίδιο και με τις προβλέψεις νομίζω μπορούμε να πούμε ότι πολλά πράγματα δεν είχαμε μπορέσει να τα προβλέψουμε, τις αλλαγές ψηφιακής οικονομίας κτλ. Και, και εσείς περιμένετε να ξαναγυρίσει ο πληθωρισμός. Ταυτόχρονα μας λέτε ότι κίνδυνοι και πλεονεκτήματα από μια τέτοια μοναδική νομισματική πολιτική είναι κίνδυνοι που ενισχύονται συν το χρόνο, αλλά και τα πλεονεκτήματα αντίστροφα μειώνονται γιατί ο κόσμο συνηθίζει αυτή τη μοναδικότητα της νομισματικής πολιτικής. Αυτό πώς το αξιολογείται. πολλές φορές οι κίνδυνοι, οι συνέπειες προκύπτουν αφού έχει περάσει το διάστημα για την δυνατότητα λήψης απόφασης. Δηλαδή βλέπουμε κινδύνους, φούσκες που μπορεί να προκύπτουν με απόκληση 12, 10, 8 μηνών. Ενώ πρέπει να λάβουμε δράση τώρα. Αυτό είναι πολύ δύσκολο. Πώς μπορούμε να το κρίνουμε αυτό και πώς μπορούμε να προστρέψουμε το βλέμμα από την πολύ επικίνδυνη νομισματική πολιτική. Όχι, κοιτάξτε, βεβαίω και κοιτούμε και το μέλλον και παρακολουθούμε την κατάσταση προσεκτικά. Μπορούμε λοιπόν να έχουμε παρά μη αναμενόμενες εξελίξεις, αλλά ταυτόχρονα αυτό μπορεί να συμβεί και ε, εάν βιαστούμε να λάβουμε αποφάσει και διαπράξουμε κάποιο σφάλμα. Πρέπει λοιπόν με κάποιο τρόπο να εξισορροπήσουμε τα πράγματα. Αυτό που άλλαξε σε σχέση με την προηγούμενη περίοδο είναι τα πολλά μέτρα πολιτικής που λήφθησαν ως απάντηση στην βαθιά χρηματοπιστωτική κρίση σε σχέση με την χρηματοοικονομική, προληπτική, μακροπροληπτική πολιτική είναι ότι μπορέσαμε να κάνουμε πιο ανθεκτικό τον τραπεζικό τομέα. Και έτσι έχουμε τη δυνατότητα να συνεχίσουμε την νομισματική πολιτική μέχρι ότου επιτύχουμε το στόχο μας. Γνωρίζουμε όμως ποιες είναι οι ελλείψεις. Και τα κενά. Την αποφάσισα. Χακμάρκ. Ναι, αλλά θέλω να ακούσω πώς τους εξετάζετε αυτούς τους κινδύνους, πώς τους βλέπετε, Πώς εξελίσσονται. Είναι οι ίδιοι με αυτούς που είχαμε πριν από ένα χρόνο, είναι ενισχυμένοι. Αλλά και τα πλεονεκτήματα. Πώς εξελίσσονται. Γιατί όσο περισσότερο έχουμε αυτή την νομισματική πολιτική, τόσο λιγότερο αποτέλεσμα θα φέρνει. Και παρά τις μεγάλες ανάγκες για ανάκαμψη το επενδυτικό κενό είναι τεράστιο. Απάντηση, ναι, η κίνδυνη πριν από ένα χρόνο ήταν υψηλότερη, αλλά προέρχονταν όχι τόσο από την οσματική μας πολιτική, όσο από τον δυνάμει αποπληθωρισμό. Τις αποπληθωριστικές τάσεις και αυτές αποτελούν κίνδυνο για τη σταθερότητα των τιμών. Και αυτό παρατηρούμε τώρα, ότι περνάμε από αυτή την κατάσταση μια νέα κατάσταση. Για τα ωφέλη εντωμεταξύ. μεταξύ για πρώτη φορά, ύστερα από πολλά χρόνια, είδαμε ένα το επίπεδο ιδιωτικών επενδύσεων που βέβαια ευνοούν τα χαμηλά επιτόκια και ασφαλώς και η ανάκαμψη με την υψηλή, υψηλή απόδοση, αποδοτικότητα ορισμένων επενδύσεων. Τα κέρδη δηλαδή ενισχύονται. Επιπλέον, ίσως θα ήταν σκοπό να ρωτούμε γιατί δεν είμαι βέβαιος ότι ε, αυτό μπορεί να συνεχιστεί ε, αυτόματα. Είπατε για την ανάκαψη, αν πρέπει να είναι αυτοσυντηρούμενη μέσω του πληθωρισμού. Αν πούμε ότι δεν είναι αυτοσυντηρούμενη ακόμη, δηλαδή χρειάζεται ακόμη την νομισματική μας πολιτική, αυτό θα έχει σε συνέπεια ότι εάν αποσύραμε την υποστήριξή μας, θα επαναρχόταν ο πληθωρισμός στα προηγούμενα επίπεδα. Ε, όλα αυτά δεν πρέπει να τα περιλάβουμε στην αξιολόγησή μας και όπως είπατε και εσείς. Πρέπει να σταθμίσουμε το κίνδυνο από την χρηματοοικονομική αποσταθεροποίηση και βέβαια τη μεσοπρόθεσμη μεσοπρόθεσμες εξελίξεις. Πρέπει να σας πω ότι μας απασχολούν και οι δύο όψεις του νομίσματος. Ευχαριστώ κύριο Πέτρος, Λίβα Περέιρα. Ευχαριστώ. Κύριε Ντράγκη, ήρθατε εδώ, πρέπει να πω, με ένα πολύ σαφές μήνυμα για την ανάγκη συνέχισης του ουσιώδους πακέτου ε, της ακολουθούμενης ε, νομισματικής πολιτικής και των κινήτων. Βεβαίως, δεν ξέρω αν η συζήτηση θα ήταν τόσο ανοιχτή αν δεν είχαν γίνει ακόμα οι γερμανικές εκλογές. Παρ' όλα αυτά αναγνωρίζουμε ότι το μήνυμα που αποστήλατε σήμερα είναι πολύ ε, σαφές. Η συμβατική ε, νομισματική πολιτική της ΕΚΤ έχει ε, επηρεάσει θετικά την ευρωπαϊκή οικονομία, ωστόσο όπως ε, έχουμε πει πολλέ φορέ η ανάκαψη είναι ανεπαρκής. ο πληθωρισμό θα μειωθεί φέτος και είμαστε ακόμα πολύ μακριά από το στόχο που έχει θεθεί για το 2019. Άρα χρειαζόμαστε ακόμη την νομισματική πολιτική, λαμβάνοντας υπόψη την κατάσταση, αλλά και τους κινδύνους. Δύο ερωτήματα για αυτούς τους ε, κινδύνους και την τρέχουσα κατάσταση. Πρώτον, προφανώς δεν θα σας ζητήσω να σχολιάσετε τα αποτελέσματα των γερμανικών εκλογών, αλλά η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα πρέπει να λάβει υπόψη της και ορισμένους πολιτικούς κινδύνους κατά τον σχεδιασμό της νομισματικής της πολιτικής. Θα λέγατε λοιπόν ότι η πολιτική αβεβαιότητα που υπάρχει αυτή τη στιγμή στη Γερμανία είναι ένας από τους λόγους που ενισχύουν την ανάγκη προ... πρόληψης κατά τον σχεδιασμό και τη διαμόρφωση της νομισματικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Και δεύτερο ερώτημα. Γνωρίζετε ότι δύο οίκοι εξολόγησης ανακοίνωσαν σημαντικές αποφάσεις τις τελευταίες ε, μέρες, που είναι η μείωση της πιστοληπτικής ικανότητας της Βρετανίας ε, βάσει του, του, ε, του Brexit βεβαίως και την ε, αναβάθμιση της Πορτογαλίας. Δεν θέλω να σχολιάσετε τις αποφάσεις οίκων αλλά θέλω να μου σχολιάσετε την κατάσταση ε, ε, η οποία έχει οδηγήσει σε αυτές τις αποφάσεις. Πώς αξιολογείτε, πώς εκτιμάτε εσείς αυτή τη στιγμή τους κινδύνους και τον αντίκτυπο του, των διαπραγματεύσεων για το Brexit στην ευρωπαϊκή οικονομία και ε, ποια είναι η γνώμη σας για την ανάκαμψη της πορτογαλικής οικονομίας. Τι στοιχεία μπορούμε να εξάγουμε από την ανάκαμψη αυτή για την συνολικά για την ευρωπαϊκή οικονομία. Ευχαριστώ. Γενικά, και όχι μόνο σε σχέση με ένα συγκεκριμένο πολιτικό συμβάν. Προφανώς και ε, λαμβάνουμε υπόψη την, ε, τις πολιτικές εξελίξεις ε, στο σχεδιασμό της νομισματικής μας πολιτικής εκτός εάν πράγματι με αντικειμενικό και άμεσο τρόπο επηρεάζεται η νομισματική μας πολιτική. Αλλιώς δεν λαμβάνουμε υπόψη, δεν υπάρχει κάποια τέτοια διάσταση. Ε, βεβαίως, ε, λαμβάνουμε ε, υπόψη μας όλα τα συμβάντα, όλα τα γεγονότα που είτε είναι πολιτικού χαρακτήρα είτε όχι, που μπορούν να επηρεάσουν την άσκηση και την υλοποίηση της νομισματικής μας πολιτικής. Όσον αφορά την αναβάθμιση της Πορτογαλίας από τη Standard Poor's, αυτή αν, αντικατοπτρίζει την ε, ε, γενική βελτίωση της κατάστασης οικονομίας της χώρας, τις μεταρρυθμίσεις που έχουν γίνει, αλλά και την εν γέννη θετική πορεία της οικονομίας Ευρωζώνης, από την οποία όλοι, όλες οι χώρες έχουν ωφεληθεί. Όπως είπα και εισαγωγικά, ε, υπάρχει ένα φαινόμενο ε, θετικού επηρεασμού, δηλαδή ε, της μίας χώρας από την άλλη. Αυτό ακριβώς το φαινόμενο παρακολουθούμε. Οι κίνδυνοι του Brexit είναι περίπλοκο να τους εκτιμήσει κανείς και θα εξαρτηθούν σε πολύ μεγάλο βαθμό από την τελική συμφωνία που θα επιτευχθεί. Αυτό που μπορούμε όμως να πούμε είναι ότι όσο περισσότερο περνά ο χρόνος, τόσο περισσότερο οι οικονομίε αρχίζουν να προσαρμόζονται στη νέα κατάσταση και όλο και περισσότερο η χρηματοστική ενδιάμεση ε, θα λαμβάνουν τις δικές τους αποφάσεις και στην ουσία θα αποφασίζουν αν θα ε, εγκατασταθούν αλλού ή όχι. Αυτό που θέλω να πω είναι ότι εφόσον υπάρχει επαρκής χρόνος και εφόσον αποφευθούν σοβαρά σφάλματα στο επίπεδο του management, η κίνδυνη αυτή είναι διαχειρίσιμη. Ευχαριστώ κύριε Ανσαντέρ. Ευχαριστώ πρόεδρε. Ευχαριστούμε πολύ κύριε πρόεδρε που είστε εδώ. Θα ήθελα να σας ρωτήσω, ποιο, να σας ζητήσω να μας πείτε ποιο είναι το μακροπρόθεσμο όραμά σας για τη ζώνη ευρώ. Καταρχήν, να σας ρωτήσω πώς μπορούμε να συνδυάσουμε επιτόκια επαρκή για να χρηματοδοτείται η οικονομία, η πραγματική οικονομία και από την άλλη μεριά ε, να εξασφαλίζουν ε, επαρκή απόδοση των καταθέσεων και των αποταμιεύσεων ενός πληθυσμού που γυράσκει. Δεύτερον, ρευστότητα των τραπεζών που δυσκολεύονται. Ερώτηση που συνδυάζεται με αυτήν του προηγούμενου συναδέλφου. Ε, το ενιαίο ταμείο εξυγίανσης που θα διαθέτει 55 δισεκατομμύρια το 2024 μόλις μπορεί να είναι πολύ περιορισμένο σε ό,τι αφορά την ικανότητα αναχρηματοδότηση των τραπεζών. Δεν πιστεύετε ότι οι, κεντρικέ οι κεντρικές τράπεζες καταρχήν και η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να στηρίξουν αυτή την ρευστότητα της ε, οποιασδήποτε τράπεζας ε, αναδιαρθρώνεται ή κατά τη διάρκεια της αναδιαρθρώσής της. Στη δεύτερη ερώτησή σας η απάντηση είναι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα δεν μπορεί να το πράξει ε, γιατί αυτό θα ισοδονομούσε με χρηματοδότηση, ε, απευθείας χρηματοδότηση. οι, ε, οι, οι, εθνικές κυβερνήσεις έχουν υποχρέωση να στηρίξουν το Ταμείο Αναδιάθρωσης Τραπεζών και εξήγιασής τους. τώρα, για τα, για τα επιτόκια, είχα, τα χαμηλά επιτόκια τόκια δημιουργούν προβλήματα και στους αποταμιευτές ε, και στους συνταξιούχους ε, που έχουν ε, ασφαλιστεί, που έχουν ασφαλιστικά συμβόλαια και για τα ταμεία σταξιοδότησης, τα εξωτικά ταμεία. Αυτοί οι δύο τελευταίοι δικαιούχοι έχουν κατά κάποιο τρόπο προσαρμοστεί, όπως και οι τράπεζες. Οι στόχοι μας είναι οι, οι, στόχοι για τα επιτόκια της ε, πολιτικής μας είναι ε, βραχυπρόθεσμοι. Οι, ε, τα επιτόκια όμως έχουν αυξηθεί με φυσιολογικό τρόπο ανεξάρτητα της πολιτικής μας. Δεν αμφιβαλώ ότι το πρόβλημα υπάρχει αλλά δεν είναι τόσο σοβαρό όσο πριν από 1,5 χρόνο. και με μια δόση ελπίδας και αισιοδοξία να πω ότι όσο βελτιώνεται η οικονομική κατάσταση, τα επιτόκια θα α, να αυξηθούν και αυτά. Και όταν μεσοπρόθεσμα ο πληθωρισμός μας φτάσει κοντά στον στόχο και είναι αυτοσυντηρούμενος τότε και η τα, δικά μας επιτόκια πολιτικής θα, είναι, θα αυξηθούν. Ποιος Φάιτσέκερ. Um, uh, Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Κύριε Πρόεδρε, κύριε Δράκη, είπατε πίστηκα ότι πρέπει να είστε πολύ προσεκτικοί τη στιγμή που μπορεί να αλλάξει η πολιτική και δεν θέλω βεβαίως να σας ε, ρωτήσω για λεπτομέρειες αυτού του χρονισμού για να μην σας φέρω σε δύσκολη θέση, αλλά τι γνώμη έχετε ως προς τα μεγέθη μακροπρόθεσμα του ισολογισμού της ΕΚΤ ο Μπεν Πενάνκι στο Jackson Hall πέρσι έλεγε ότι εν όλο οι κεντρικέ τράπεζε θα πρέπει να έχουν όλο και μεγαλύτερο ισολογισμό με πολύ εύστοχα επιχειρήματα. Αλλά υπήρχε και ένα αρνητικό όταν επεσήμανε ότι υπάρχει και ο χρηματοοικονομικός κίνδυνος και μάλιστα ανέφερε ότι για τις ΗΠΑ δεν είναι μεγάλος, αλλά η Ευρωζώνη κινδυνεύει περισσότερο. Έτσι λοιπόν με δεδομένη αυτή τη συζήτηση και μακροπρόθεσμα θέλω να μου πείτε ποια είναι η γνώμη σας. Όταν ε, η νομισματική κατάσταση, ο ισολογισμός της ΕΚΤ τι μεγέθη πρέπει να έχει. Και κάτι ακόμη για το σύστημα εξυγίανσης CCP που αναφέρατε και πέρσι και εσείς στις συζητήσεις και είχατε πει ότι οι κεντρικές τράπεζες έχουν σημαντικό ρόλο όταν ε, οι, οι μεγάλες τράπεζες ε, έχουν πρόβλημα, οι CCPs, τότε μήπως θα έπρεπε να κοιτάξουμε την προσέγγιση των, τη ρυθμιστική όταν είναι πιο, πιο συστημικές ακόμη οι CCPs από ορισμένε μεγάλες τράπεζες. Η, η θέση αυτή μπορεί να στέκει. Οι κεντρικές τράπεζες μήπως έχουν πιο μεροληπτική στάση και σχέση με ορισμένους μεγάλους παράγοντες της αγοράς. Μήπως χρειάζεται ένα ενιαίο σύστημα εξυγίανσης και ανάκτησης για τις που έχουν μεγάλη σημασία ε, διασυνοριακά, αντίστοιχα με αυτά που έχουμε κάνει δηλαδή για τις τράπεζες. Απάντηση θα απαντήσω στη δεύτερη ερώτηση σας πρώτα. θα είδατε ότι η τροποποίηση του άρθρου 22 προς αυτή την κατεύθυνση πηγαίνει μαζί με την ε, αναθεωρημένη πρόταση Επιτροπής. Υπάρχουν κάποιες δεσμευτικές εξουσίες για την Κεντρική Τράπεζα έκδοση, που σημαίνουν αναγνώριση του, ε, της ΕΣΥΠΗ σε μια χώρα τις δυνατότητες επανεγκατάστασης ή μετεγκατάστασης και κάποιες ρυθμιστικές δραστηριότητες. Η Κεντρική Τράπεζα Έκδοσης δεν μπορεί να είναι απευθείας επιβλέπουσα της CCP's ή των CCP's. Και αυτές θα πρέπει να υπάγονται σε διαφορετικό εποπτικό σύστημα. Αυτό σημαίνει όταν λέτε ότι και εσείς ότι ειδικά όταν είναι συστημικές αυτές και εδώ ακριβώς θέλουμε η... Εδώ είναι ακριβώς που θέλουμε θέλουμε ακριβώς αυτήν την εποπτεία για τους κεντρικούς αντισυμβαλόμενους. Για την πρώτη σας ερώτηση τώρα, ο ισολογισμό της ΕΚΤ, πόσο μεγάλος μπορεί να είναι. Μα αυτό εξαρτάται από τα μεγέθη της οικονομίας και την επίτευξη των στόχων, ή κατά πόσον έχουν επιτευχθεί οι στόχοι. Έχουμε σημειώσει ότι το μέγεθος του ισολογισμού μπορεί να είναι νομισμα... μέσων εργαλείων νομισματικής πολιτικής. Εμείς το κάναμε πρώτο αυτό. Και αυτό είναι και το νόημα όλες τις προσπάθειες. Δεν λέμε αν πρέπει να υπάρχει ένα επίπεδο συγκεκριμένο επιτοκίων πέραν των οποίων δεν πρέπει να προχωρήσουμε ή χαμηλότερο, αντίστοιχα, ή πιο πριν που ήταν και αρνητικά. Δηλαδή δεν υπάρχει κάποιος προκαθορισμένος όγκος. Απλώς λέμε και ξέρουμε ότι είναι ένα εργαλείο που πρέπει να είναι διαμορφωμένο, διαπαθμισμένο, έτσι ώστε να εξυπηρετεί το στόχο μας. Και ξέρουμε αν μπορεί να τον εξυπηρετήσει ή αν μας απομακρύνει από το στόχο μας και αν η σύγκληση είναι δυνατή ή όχι. Ωστόσο, τα μεγέθη του ισολογισμού είναι ένα μέσο, ένα εργαλείο. Και θα εξαρτηθεί βεβαίω η επιτυχία μας από το τι κάνουμε και από τα άλλα μέσα που έχουμε στη θέση μας. Ήδη είναι πολύ δύσκολο να αξιολογήσει κανείς ένα πρότυπο μεγέθους το οποίο θα ίσχυε για τους πάντες και ανά πάσα χρονική στιγμή. Πολύ δύσκολο αυτό. Ευχαριστώ κύριο Λουκέ. Μάλλον έφυγε γιατί δεν ήταν τόσο τέλεια η ερωτήση για την τελική απάντηση. Οι τελικές απαντήσεις μάλλον. Θα του δώσετε γραπτός ο κύριος Ευχαριστώ. Εδώ είμαι και θέλω να θέσω το ερώτημά μου στα Ολλανδικά. Καλησπέρα. Θέλω να σας ρωτήσω κάτι που σχετίζεται με την ανακοίνωση της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας. Είναι σημαντικό εργαλείο που έχετε στα χέρια σας ε, προκειμένου να αντιμετωπίζετε το ζήτημα του πληθυσμού και να επηρεάζετε τις ε, χρηματαγορές. είναι σημαντικό η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα να είναι ένας, ένα θεσμικό όργανο διαφανές. Υπάρχουν λοιπόν, υπάρχει λοιπόν κάποια συγκεκριμένη ανακοίνωση σχετικά με τα προγράμματα κινήτρων. Γιατί ακούγεται πολύ συχνά η κατηγορία ότι υπάρχει έλλειψη διαφάνειας, κάτι που επηρεάζει αρνητικά την οικονομική σταθερότητα. Γιατί ακούγεται, ακούγονται φήμες ότι θα υπάρξουν αυξήσεις Ενώ από την άλλη πλευρά ε, ε, ε, υπάρχει άποψη ότι κάτι τέτοιο δεν πρέπει να γίνει στο πλαίσιο στο πλαίσιο στο οποίο βρισκόμαστε σήμερα και ακόμα δεν έχει ξεπεραστεί πλήρως η οικονομική κρίση. Δεν θέλω βεβαίως να συγκρίνω την Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα με την Fed, διότι έχουν διαφορετικές αρμοδιότητες. Θέλω όμως να σας ρωτήσω γιατί δεν χρησιμοποιείτε αυτό το εργαλείο ε, των, ε, των ανακοινώσεων ε, με έναν πιο αποτελεσματικό τρόπο. Ρωτάτε αν μπορούμε να, να βελτιώσουμε την επικοινωνική μας ε, στάση και πολιτική. Φυσικά, περιθώρια βελτίωσης υπάρχουν πάντοτε. Μέχρι στιγμής, ωστόσο, νομίζω ότι η αίσθηση που έχω είναι ότι η επικοινωνική στρατηγική της ΕΚΤ είναι αρκετά ε, αποτελεσματική σε πολλές περιστάσεις. Έχουμε μάλιστα διάφορους διάβλους ε, επικοινωνίας. Για παράδειγμα, ε, το, το, το, το δελτίο τύπου, οι συνεντεύξεις τύπου, οι ομιλίες των μελών του Διοικητικού Συμβουλίου μας. Από αυτή την άποψη λοιπόν νομίζω ότι η επικοινωνική μας τακτική είναι αρκετά στιβαρή και νομίζω ότι η, η αίσθηση που έχω, βεβαίως μεροληπτό εν μέρη, ε, είναι ότι η συγκεκριμένη ε, ανακοίνωση επέτυχε το στόχο της. Αν ε, θέλετε να εξετάσουμε τους, ε, το, επόμενο διάστημα, το διάστημα των επόμενων μηνών, νομίζω ότι το Διοικητικό Συμβούλιο της ε, ΕΚΤ έχει αφιερώσει τον απαραίτητο χρόνο προτού εισέλθουμε σε αυτή τη νέα φάση. Και πιθανόν στην επόμενη συνάντηση για την νομισματική πολιτική, το, το φθινόπωρο, ε, θα συζητήσουμε ε, αυτό το, το ζήτημα των, ε, της κατάστασης της, της ασκούμενης νομισματικής πολιτικής για τις επόμενους μήνες. Θα μου πείτε, γιατί περίμενε το, γιατί περίμενε το Διοικητικό Συμβούλιο τον Οκτώβριο να γίνει αυτό. Δεν μπορούσε να το έχει κάνει και τον Ιούνιο. Είναι ένα θέμα που το έχουμε συζητήσει και εμείς, πρέπει να σας πω. Ωστόσο, η αβεβαιότητα που καθημερινά ε, υπάρχει από διάφορες εξελίξεις και εκπλήξεις είναι τόσο μεγάλη που μας οδήγησε ε, και οδήγησε ιδίω τα κράτη-μέλη στην, ε, στην άποψη ότι όσο περισσότερες πληροφορίες έχουμε στα χέρια μας τόσο καλύτερα θα τροφοδοτηθούν και οι συζητήσεις που θα έχουμε. Ε, και βεβαίως στο πλαίσιο ε, αυτούς της, της επικοινωνικής υπάρχει και αυτό το monitor, αυτός ο διάλογος εδώ με το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Βεβαίως λέει ο κύριος ε, Ντράγκη. Ευχαριστώ. Ο κύριος Τάγκ. Όταν ε, σας ε, ε, επισκεφτήκαμε η αποστολή της Επιτροπής μας ε, ε συζητήσαμε πάρα πολλά ενδιαφέροντα ε, ζητήματα. Η συζήτηση ήταν πολύ ενδιαφέρουσα. Ε, ποια είναι η γνώμη σας λοιπόν για την προσαρμογή της Ευρωζώνης μεσοπρόθεσμα. Γιατί Αντιμετωπίζουμε αυτό το πρόβλημα στην Ευρωζώνη. Υπάρχει ένα μείγμα νομισματικής και δημοσιονομικής πολιτικής. Είναι πρόκληση αυτό. Αλλά πώς ε, αξιολογείται και τις εξελίξεις που υπάρχουν στις ορισμένες χώρες, ιδίως ε, ε, εκείνες τις χώρες όπου υπάρχει πλεόνασμα των τρέχουσων συναλλαγών, βλέπετε στην Γερμανία αλλά και σε άλλες χώρες παρόμοιες οι μισθοί δεν αυξάνονται, κάτι που δεν ε, βοηθά την, ε, την, ε, τη σύγκληση και την προσαρμογή. Και μάλιστα η κατάσταση επιτείνεται ακόμα περισσότερο από το γεγονός ότι δεν έχουν σχηματιστεί ακόμα κυβερνήσεις στις χώρες αυτές. Ε, εσείς ποια μέτρα πιστεύετε ότι πρέπει να ληφθούν προκειμένου να ενισχυθεί και να βελτιωθεί η προσαρμογή στις χώρες αυτές. Πράγματι, ε, ε, μισθολογικές εξελίξεις αυτή τη στιγμή ε, βρίσκονται χαμηλότερα από ό,τι ε, είχαμε συνηθίσει στο παρελθόν σε αυτή τη φάση του κύκλου της οικονομίας. Υπάρχουν πολλοί λόγοι. Ε, οι περισσότεροι από αυτούς σχετίζονται με τη λειτουργία της αγοράς εργασίας. Θα σας παραθέσω κάποιους από αυτούς τους λόγους. Πρώτον, βγαίνουμε από μια παρατεταμένη περίοδο δυσκολιών στην ε, αγορά εργασίας. Υπάρχει λοιπόν μια παρακαταθήκη αυτή τη στιγμή του παρελθόντος, η οποία μετουσιώνεται αυτή τη στιγμή σε μια κατάσταση στην αγορά εργασίας, όπου η ανεργία είναι πιθανότατα υψηλότερη από, από ό,τι λένε τα επίσημα στοιχεία. Τα γνωστά στοιχεία U6, όπου πολλοί απασχολούμενοι, εργαζόμενοι, έχουν συμβάσεις ορισμένου χρόνου ή βρίσκονται σε καταστάσεις, σε, σε, σε, σχέσεις εργασίας χαμηλής ποιότητας, κάτι που δεν ε, βεβαίως βοηθά στην αύξηση των μισθών. Επίσης, ο χαρακτήρας αυτών των συμβάσεων ε, ορισμένου χρόνου ε, αποτελεί θέμα που απασχολεί και τα συνδικάτα. Τα συνδικάτα όμως έχουν θέσει πιο πολύ στο επίκεντρο της προσοχή τους όχι τόσο την αύξηση των μισθών όσο τη σταθερότητα των σχέσεων εργασίας. Ένας άλλος λόγος είναι το γεγονός ότι υπάρχει μια παρακαταθήκη. Κατά τη διαπραγμάτευση λοιπόν για τα μισθολογικά ζητήματα αυτές οι συζητήσεις έχουν στραμμένο το, το, το βλέμμα τους στο παρελθόν, στο ποιος, πώς, πως που, που κινούνταν ο πληθωρισμός τα τελευταία 3-4 χρόνια και έτσι οι αυξήσεις που ζητούνται από τα συνδικάτα είναι χαμηλότερες και δεν αντιστοιχούν στον τρέχοντα πληθωρισμό. Επίσης, κάτι που δεν συνδέεται βεβαίως με την αγορά εργασίας είναι το χαμηλό επίπεδο της παραγωγικότητας. Η παραγωγικότητα είναι ε, χαμηλή ε, σε, σε, όλους σχεδόν τους ε, τομείς, εκτός από τον εξαγωγικό τομέα βεβαίως. Όλοι αυτοί οι παράγοντες λοιπόν συντελούν στο να κρατιούνται οι ονομαστικοί μισθοί σε χαμηλά επίπεδα. Αυτό που εμείς πρέπει να κάνουμε είναι να επιδείξουμε υπομονή. Διότι πιστεύουμε ότι ο πληθωρισμός μέσω και μακροπρόθεσμα θα υπηρετήσει τους στόχους που έχουμε θέσει, διότι τα οικονομικά στοιχεία ε, θα βελτιωθούν, κάτι που θα οδηγήσει και σε κλείσιμο ε, του, του, του, του χάσματος μεταξύ αποδοτικότητας και μισθών, αλλά πρέπει να είμαστε υπομονητικοί, διότι αυτά τα πράγματα δεν μπορεί να γίνονται αυτόματα. Και γι' αυτό, εκτό από υπομονή, πρέπει να επιδεικνύουμε και επιμονή. Δεν μπορούμε να προβούμε σε βεβαιασμένε κινήσει, Πρέπει να είμαστε πολύ προσεκτικοί σε αυτά που κάνουμε. Ευχαριστώ. Ο κύριος Κίρτσο έχει το λόγο. Thank you, uh, Πρόεδρε Ντράγκη, και οι ελληνικές εταιρείε όσο και το ελληνικό δημόσιο ε, επιθυμούν να ενταχθούν στο πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας για να καλύψουν τις χρηματοδοτικές τους ανάγκες ε, και να μειώσουν το κόστος δανειοδότησης. Ε, πότε και υπό ποιες συνθήκες θα μπορούσε να επιτευχθεί αυτή η θετική εξέλιξη. Και δεύτερον, σκέφτεστε να αναλάβετε κάποια καινούργια πρωτοβουλία προκειμένου να βοηθήσετε τις ε, ελληνικές τράπεζες να ξεπεράσουν τα αποτέλεσμα της κρίσης του 2015. Τα, τους τελευταίους μήνες ο τραπεζικός τομέας στην Ελλάδα δέχεται όλο και περισσότερες ε, πιέσεις από το Διεθνές Νομισματικό Τομέα ε, που ενδεχομένως τίνουν στο να οδηγήσουν σε μια καινούρια ανακεφαλαιοποίηση των τραπεζών στην Ελλάδα. Πώς μπορούμε να το αντιμετωπίσουμε. Ο κ. Δράγκη. Να σας απαντήσω τη δεύτερη ερώτηση πρώτα. Ε, οι αποφάσεις μας λαμβάνονται σε πλήρη ανεξαρτησία. Το, οι αποφάσεις του SSM μάλλον είναι τελείως ανεξάρτητες. Ε, του χρόνου θα γίνει ένα stress test ε, για τις τράπεζες και κατά βάση ο SSM έστειλε και μια επιστολή στο Διεθνές Ταμείο για αυτό το stress test που θα διοργανώσει του χρόνου. Σε ό,τι αφορά την πρώτη ερώτηση θα μπορούσατε να μου επαναλάβετε την ερώτηση γιατί δεν την κατάλαβα. Χωρίς μικρόφωνο αυτή τη στιγμή ο κ. Κίτσος. και οι ελληνικές ιδιωτικές εταιρείες και το κράτος ε, επιθυμούν ε, να ενταχθούν στο πρόγραμμα αγοράς περιουσιακών στοιχείων της Ευρωπαϊκής Κεντρικής Τράπεζας προκειμένου να καλύψουν τις ε, χρηματοδοτικές ανάγκες και να μειώσουν το κόστος δανεισμού. Πότε και υπό ποιε συνθήκες θα μπορούσε να προκύψει αυτή η θετική εξέλιξη. Ο κ. Δράγκη. Όπως ξέρετε και φαντάζεστε, έχω ρωτηθεί για το θέμα αυτό πολλές φορές. Το σημείο κλειδί είναι ότι η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα πρέπει να κάνει ε, ε, μια αξιολόγηση ε, του βιώσιμου του χρέους. Και αυτή η αξιολόγηση θα είναι δυνατή μόλις έχουμε αρκετές πληροφορίες και σαφείς πληροφορίες για, το, τα μέτρα για το χρέος Ελλάδος που θα λάβει το Eurogroup και τα κράτη-μέλη. Η αξιολόγηση του βιώσιμου του χρέους θα πρέπει να λάβει υπόψη και όλους τους ε, εξωτερικούς κινδύνους. Τότε η Ευρωπαϊκή Κεντρική Τράπεζα θα μπορούσε να συζητήσει το θέμα της ένταξης της Ελλάδας στο πρόγραμμα ε, ποσοτικής χαλάρωσης. Σας ευχαριστώ. Συναρπαστικός νομισματικός διάλογος. Ευχαριστώ τον πρόεδρο Ντράγκη και όλους τους συναδέλφους που συνέβαλαν στη συζήτηση. Θα συνεχιστεί και βεβαίως προσβλέπουμε στις προσεχείς αποφάσεις για την νοσματική πολιτική της ΕΚΤ. Σας ευχαριστώ όλους. Παρακαλώ, αγαπητοί συνάδελφοι, καθίστε. Για να περάσουμε στο σημείο 3 της ημερήσιας διάταξης, ανακοινώσει του Πρόεδρου. Όπως έχει συμβεί και σε προηγούμενες χρονιές, αντιπρόσωποι των Εθνικών Κοινοβουλίων θα μας επισκεφθούν στις 10 Οκτωβρίου, 3 με 4.30 πριν από την ψηφοφορία στην Επιτροπή της δεύτερης έκθεσης πρωτοβουλίας για το εξάμεινο, προκειμένου να συζητήσουμε διαρθρωτικές μεταρρυθμίσεις και ε, χρηματοοικονομικές επιλογές που θα υλοποιηθούν στις χώρες, τους δημοσιονομικές μάλλον επιλογές. Φέτος ε, έχουμε και άλλη ανταλλαγή απόψεων που ξεκινάει μέσα μετά τα 4.30 την ίδια μέρα για πρόταση για κοινό εταιρικό ε, συντελεστή, φορολογικό συντελεστή ε, και πρόταση για ένα κοινό ενοποιημένο φορολογικό συντελεστή. Δεδομένου ότι έχουμε εκφραστεί διάφορε τέτοιε γνώμε από διάφορα εθνικά κοινοβούλια, η Επιτροπή θέλει να συζητήσει με εκπροσώπου ε, των Εθνικών Κοινοβουλίων ε, των ευκαιριών αυτών για μια κοινή λοιπόν φορολογική βάση. Και θα έχετε ίσως παρατηρήσει, θα έχετε ακούσει ότι στους διαλόγους 7 και 12 Σεπτεμβρίου επετεύχθη τελικά γενική πολιτική συμφωνία μεταξύ των συνομοθετών στον τριμερή διάλογο σε διάφορα θέματα, βασικά θέματα εκρεμεί όπως ο προϋπολογισμός, η διακυβέρνηση, η τιμολόγηση, προσθετικότητα και διάφορα άλλα σημαντικά θέματα. υποστηρίζει την συμφωνία αυτή το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο βεβαίω. αν και θα πρέπει να την εγκρίνει ρητά, να εκφράσει γνώμη, αλλά νομίζω ότι μπορούμε και με την έγκριση της πρότασης του ΕΦΣΥ να πούμε ότι και το Κοινοβούλιο και το Συμβούλιο συγγνώμη, φάνηκε σε έναν τελικό τριμερή διάλογο διτεθειμένο να ολοκληρώσει όλη την ε, συμφωνία και μπορούμε να ολοκληρώσουμε την ε, νομοθετική αυτή διαδικασία το του δυνατό έτσι ώστε να συμβάλλουμε στην ε, παράταση και βελτίωση, επέκταση, παράταση και βελτίωση του νομοθετικού σχεδίου. Πρακτικά επίσης, 30-31 Αυγούστου 4 Σεπτεμβρίου. Εάν δεν υπάρχουν αντιρρήσεις θα εγκρίνουμε. Και σας ευχαριστώ και πάμε στο σημείο 6. Εκτέταση τροπολογιών στην έκθεση του κυρίου Χόκμορκ για την ε, κατάταξη των μη εξασφαλισμένων χρωστικών μέσα στην πληγευτική ιεραρχία. Δεν θα ψηφίσουμε, όπως ξέρετε, μετά τη συζήτηση αλλά θα ακούσουμε πρώτα τα σχόλια του εισηγητή για τις διάφορες τροπολογίες. Ψηφοφορία θα γίνει ούτως ή Μετά στα άλλα θέματα, γι' αυτό μην αποχωρήσετε, γιατί προβλέπονται ακόμη δύο θέματα προς ψηφοφορία. Έχετε το λόγο κύριε Χοκμάρκ. Ευχαριστώ πολύ πρόεδρε. Καλώς ορίζω. Ε, όλες τις ε, τροπολογίες που έχουν κατατεθεί βεβαίως Δύσκολα νομίζω μπορεί να εντοπίσει κανείς σοβαρές πολιτικές διαφωνίες, απλώς πρόκειται για διευκρινήσεις, ε, αναζήτηση σαφήνειας ή πιο συνεπούς κειμένου. Μερικές φορές όμως η συνέπεια στο κείμενο μπορεί να μην είναι ε, σύμφωνη με άλλες τροπολογίες, ακόμη και αν τευκόλυνει τη διαφάνεια. Ε, αυτό πρέπει να ξέρει κανείς στα πράγματα στα τεχνικά τους σημεία για να το επισημάνει. Επίσης έχω, ή έχω σκοπό να διανύμω συμβαστικές τροπολογίες είτε αύριο είτε μεθαύριο, προκειμένου να διευκολύνουμε αυτή την προσπάθεια, να ανταποκριθούμε δηλαδή σε όλες ε, τις ανησυχίες και τα μελήματα, χωρίς όμως να υπονομεύουμε τη σαφήνεια και την συνοχή του κειμένου. Και πάνω απ' όλα, κύριος στόχος μας είναι η σαφήνεια, δηλαδή η ιεράρχηση να είναι σαφής. Έτσι λοιπόν κάποιες τροπολογίες που μπορεί να μην αλλάζουν σοβαρά το κείμενο, μπορεί να είναι αρκετά συναφείς. Θα ήθελα να επισημάνω ότι μπορούν να αποδεκτέ ε, διαφορέ σε εθνικέ ε, νομοθεσίε προκειμένου να γίνουν σεβαστέ ή ήδη υφιστάμενε στα κράτη-μέλη νομοθεσίε. Εθνικέ νομοθεσίε. Ωστόσο, θα ήθελα να επισημάνω ότι θέλω να διατηρηθεί αυτή η δυνατότητα ε, για τις εθνικές δικαιοδοσίες που έχουν ήδη ρυθμίσει τα θέματα αυτά. Για το θέμα της ε, μετάβασης, τη ρήτρα grandfathering, πρέπει επίσης να βρούμε μία λύση διαφανή, προβλέψιμη για όλους τους εμπλεκόμενους παράγοντες της αγορές. Την επόμενη εβδομάδα θα έχουμε συνεδρίες των σκιωδών κατά την οποία ελπίζω ότι θα μπορέσουμε να καταλήξουμε σε συμφωνία στα περισσότερα θέματα, όπως και να έχει. Δεν πιστεύω ότι μπορεί κανείς να αισθάνεται απογοητευμένος από το αποτέλεσμα, γιατί οι διαφορές δεν οδηγούν προς, προς μεγάλη διαφοροποίηση. Ευχαριστώ πολύ, λέω Ευχαριστούμε για τη δουλειά σας. Δεν νομίζω ότι θα είναι κανείς απογοητευμένος αλλά πάνω απ' όλα θα έχουμε την ευκαιρία όλοι να ψηφίσουμε, γιατί έχει προεξαγγελθεί για την ε, Ολομελία του Οκτωβρίου το θέμα αυτό. Ας είμαστε αισιόδοξοι λοιπόν. Συζητούμε με την κυρία Σίλβα Περέιρα πρώτα, τους Αριστές Δημοκράτες. Τον κύριο Σίλβα Περέιρα. Ευχαριστώ. Πρόεδρε. Να σας υπενθυμίσω καταρχήν ότι η πολιτική μας ομάδα εξ αρχής ε, επιστήριξε την ταχεία διεκπαιρέωση του θέματος ε, του φακέλου αυτού. Χρειάζεται να προχωρήσουμε γρήγορα και βαίνουμε προς τη σωστή κατεύθυνση εν γέννη. Παρ' όλα αυτά, πρέπει να συζητήσουμε την έκθεση. Ε, καλωσορίζω την, το καινούριο χρονοδιάγραμμα συζήτησης. Ως εισηγητής θεωρώ ότι το γεγονό ότι έχουμε 69 τροπολογίες δεν σημαίνει απαραίτητα ότι υφίσταται κάποια βαθιά πολιτική διαφωνία που να είναι δυσεπίλητη. Είμαστε κι εμείς αισιόδοξοι σε ό,τι αφορά τις συζητήσεις που θα γίνουν την ερχόμενη εβδομάδα. Να υπογραμμίσω εντάχει μερικά ζητήματα που είναι σημαντικά για μας σε τροπολογίες που υπέβαλα εκ μέρους ομάδας μου. Καταρχήν, για την πατρογονική ρήτρα, είναι πολύ σημαντικό να δώσουμε το μήνυμα ότι το στόκ του υπάρχοντος χρέους θα υπαχθεί σε αυτή την ρήτρα όλα τα μέσα τα οποία έχουν εκδοθεί προ της ε, ε, έκδοση των κριτήριων επιλεξιμότητας θα πρέπει να ενταχθούν. Ε, μετά, η σημαντική οριμότητα θα πρέπει να είναι τουλάχιστον ενό έτους σε αυτά τα μέσα τα οποία εκδίδονται. Ε, τουλάχιστον ένα χρόνο Λοιπόν, ε, έτσι κι αλλιώς αυτό προέλεπαν οι ελάχιστες απαιτήσεις ιδίων κεφαλαίων, η ΕΜΡΕΛ. Ε, πρέπει να φτάσουμε τουλάχιστον λοιπόν στο επίπεδο των MR, ε, MREL. Η, η οδηγία θα πρέπει επίσης να είναι με την φύλαξη ε, οποιασδήποτε εθνικής διάταξης, ε, ε, προτιμησιακής διάταξης για τους καταθέτες. Έτσι, ε, δεν μπορεί να υπερτεθεί έναντι των εθνικών επιλογών και προτιμήσεων. Σε ό,τι διαφορά αφορά το θέμα του κατά πόσον τα κράτη-μέλη θα πρέπει να επιτρέπεται να τρέξουν πιο γρήγορα, αν το επιθυμούν, Πιστεύουμε ότι ναι, θα έπρεπε να τους επιτραπεί. Ε, θα μπορούσαν, αν το επιθυμούν, να ε, εισάγουν το σύστημα πιο νωρίς. Σε ό,τι διαφορά την έναρξη ισχύω, πιστεύουμε ότι μια γρήγορη έναρξη ισχύω θα ήταν χρήσιμη. Οπότε στηρίζουμε μια περίοδο δύο μηνών. Αυτές είναι οι βασικές μας προτάσεις τροπολογιών και είμαστε, σε, και είμαστε πρόθυμοι να τις συζητήσουμε με τις άλλες πολιτικές ομάδες. Ευχαριστώ. Επόμενος ομιλητής για το ECR, ο κύριος Καμάλ. Ευχαριστώ. Ευχαριστούμε τον εισηγητή και τους ε, άλλου σκιώδει. Νομίζω ότι οι συνεδρίες που είχαμε μέχρι στιγμή ήταν επικοδομητικές και ε, ε, χαρακτηρίστηκαν από πνεύμα συνεργασία και όχι, και όχι διαφωνία. Εμεί υποστηρίζουμε τι τροπολογίε του εισηγητέ για. Ως, ιδίως όσον αφορά την, το χρέος υψηλής προτεραιότητας. Απλά δεν θα πρέπει οι τροπολογίες αυτές να έρχονται σε αντίθεση με εθνικούς κανόνες ε, για την αφαιρεγγιότητα ε, και είναι πολύ σημαντικό επίσης να δοθεί αυτή η νομική βεβαιότητα, κάτι που βεβαίως πιστεύω ότι συνάδει, συνάδει με την έκθεση του συγητή. και θα ήθελα να ακούσω και τις απόψεις των άλλων ε, πολιτικών ομάδων. Βεβαίως θα ήθελα να μας υποστηρίξουν σε αυτό, αλλά θέλω κυρίως να ακούσω τις απόψεις τους. Όσον αφορά την, τον προαιρετικό χαρακτήρα ε, ε, ε, της, ε, την, την τροπολογία των πρασίνων, σε εκείνη αναφέρομαι, εμεί διαφωνούμε. Όσον αφορά τις τροπολογίες των άλλων χωρών, ομάδων, το να νομίζω ότι πρέπει να υπάρχει κάποια ευελιξία ε, όσον αφορά τους κανόνες, αλλά μόνο κατ' εξαίρεση, για να μην υπάρξει υπερβολικός ε, κατακαιρματισμός. Εγώ ε, γενικά συμφωνούσα με την περίοδο των 12, μηνών. Ε, απλώς ε, φαίνεται ότι υπάρχει μια τροπολογία, κάποια στοιχεία στην έκθεση μάλλον, που έρχονται σε αντίθεση με το πρότυπο TILAC. Επίσης, είμαι επιφυλακτικός με την ε, προτίμηση εναντί καταθετών ε, χρέος, γιατί αυτό ενδεχομένως να στρεβλώσει την, ε, την, την αγορά. αλλά αυτά είχα να πω ως σχόλια. Περιμένω να ακούσω και τις απόψεις των άλλων. Ο κύριος Κορνιγέ από τους Φιλελευθέρους έχει το λόγο. Δεν είναι εδώ. Δεν υπάρχει εκπρόσωπος των Φιλελευθέρων. Ωραία. Γκουε η κυρία Ματίας εκ μέρους του κυρίου Ντεμάζη που, πλέον εξελέγει στο Bundestag ε, Μαρίζα. Ευχαριστώ Ρομπέρτο. Ξέρεις ότι δεν είμαι σκιώδης, αλλά δυστυχώς ο Φάμπιο δεν μπορεί να είναι σήμερα εδώ, καθώς εξελέγει βουλευτής του Γερμανικού Κοινοβουλίου. Έχει πολύ σημαντικό λόγο δηλαδή που ε, απουσιάζει. Όπως και να έχει, θα προσπαθήσω να χρησιμοποιήσω τις σημειώσεις που μου έχει δώσει και να υποβάλω τα σχόλιά μου στον εισηγητή. Τον ευχαριστούμε λοιπόν για την επικοδομητική του στάση. Έχουμε υποβάλει κάποιες βασικές σημαντικές τροπολογίες που θεωρούμε ότι θα καταστήσουν το σύστημα ε, διάσωσης με ίδια μέσα πιο αξιόπιστο. Θεωρούμε ότι ε, οι τράπεζες εξακολουθούν να μην έχουν επαρκή κεφαλαιοποίηση. Ε, θεωρούμε ότι εξακολουθεί να υπάρχει η, μια ε, αντίληψη η οποία ε, αναφέρει ότι κάποιες τράπεζες είναι υπερβολικά μεγάλες για να αποτύχουν. Κάτι που μπορεί να δημιουργήσει μεγάλα προβλήματα. Οι τράπεζες λοιπόν έχουν στοιχεία παθητικού ε, που θα πρέπει να μπορούν να ε, καλύπτονται σε περίπτωση ανάγκης. Γι' αυτό και χρειάζεται μια σαφής ιεράρχηση και συμφωνούμε με τον εισηγητή ότι επί της ουσίας όλα το, όλο το χρέος θα πρέπει να είναι ε, διασώσιμο με ίδια μέσα. Αυτό ε, έχουμε δει όλοι ε, αναφορές στον τύπο ο, βάσει των οποίων επενδυτές ασκούν ε, αγωγές κατά ε, κρατικών φορέων. Χρειαζόμαστε βεβαιότητα. Γι' αυτό και θεωρούμε ότι ε, πρέπει να εξασφαλιστεί ότι το χρέος θα είναι χαμηλότερης προτεραιότητας έναντι όλων των άλλων των στοιχείων παθητικού. Δεν συμφωνούμε με τον εισηγητή ότι οι τράπεζες θα πρέπει να επιτρέπεται να εκδίδουν όλα τα είδη χρέους, γιατί αυτό θα περιβλέξει τα πράγματα και θα ενισχύσει την αδιαφάνεια. Και όπως και άλλες πολιτικές ομάδες δεν θέλουμε να διαγραφεί η ελάχιστη διάρκεια ενός έτους όπως προτείνεται στην τροπολογία 20. Επίσης πιστεύουμε ότι ε, το χρέος δεν πρέπει να πωλείται σε ε, μη εγκεκριμένου επενδυτέ και, να υπάρχει σύγχυση μεταξύ αυτών των επενδυτών και των καταθετών. Επίση, για τι πατρογονικέ ρήτρε πιστεύουμε ότι πρέπει να ισχύσουν σε περιπτώσει όπου τα κράτη-μέλη έχουν επιλέξει εναλλακτικό σύστημα προ την ε, συμβατική χαμηλή προτεραιότητα. Παρ' όλα αυτά, προσβλέπουμε και στι από εδώ και πέρα συζητήσει που θα έχουμε με τον εισηγητή. Ευχαριστώ κύριο Λάμπερτς. Πού το μαντέψατε ότι φέτος θα με ο Ερνέστ. Μπορεί να μην είναι τόσο καλά τα ισπανικά μου, αλλά τα καταφέρνω. Θα το διαβάσω όσο πιο ζωντανά γίνεται για να μην αποκοιμηθείτε. Αν βαρεθείτε παρακαλώ πολύ κάντε μου ένα νόημα με το χέρι, έτσι μια ευγενική χειρονομία. Καταρχήν, Γκιουνά, εσύ και εγώ, η ιστορία αγάπη αυτή έρχεται από πολύ μακριά, από πολύ πίσω. Δεν ξέρω αν θα πρέπει να το πω, Τέλο πάντων. Σε συγχαίρουμε που ευθυγραμμίστηκες με το Συμβούλιο. Αυτό, θα, αυτό μας οδηγεί σε μια συμφωνία σε πρώτη ανάγνωση. Ε, το TLAC, τα πρότυπα του TLAC είναι πολύ σημαντικά και χαιρόμαστε που αναφέρεις αυτά. Έχουμε τρία θέματα που θα ήθελα να λάβεις υπόψη σου. Πρώτον, να το διαβάσω γιατί δεν είμαι σίγουρος ότι καταλαβαίνω και πολύ καλά. Όλες οι μη εμπορεύσιμες, ε, όλα τα στοιχεία θα πρέπει να έχουν ε, ε προτεραιότητα και αυτό έρχεται σε αντίθεση με αυτό που ελέγχθη προηγουμένως. Ε, τα στοιχεία αυτά θα πρέπει να χρησιμοποιηθούν πιο νωρίς από τα άλλα γιατί έτσι το σύστημα θα γίνει πιο αποτελεσματικό και θα επιταχυνθεί η εξυγίανση. Κάτι πραγματικά χρειάζεται. Δεύτερον, θέλουμε να απαιτείται όλες οι απαιτήσει σε εμπορεύσιμο χρέος να ε, ε, εμπίπτουν σε κάποια πρότυπα τα οποία δεν καταλαβαίνω, θα μου το εξηγήσει κάποιος. Ε, και τρίτον, ε, μια και έχουμε μια νέα κατηγορία μέσων που δημιουργούνται με την DRRB και τώρα, σε, από πλευρά θα πρέπει να θεωρούνται ως ε, σύνθετα όργανα μέσα και θεωρούμε ότι οι διατάξει της Μύφιτ για τη σύγκρουση συμφερόντων θα πρέπει να ισχύουν για την πώληση τέτοιων μέσων. Αυτά μου ζήτησε η ομάδα μου να πω. Ελπίζω να είστε ακόμα ξύπνοι και νομίζω ότι μπορούμε να χρησιμοποιήσουμε το χρόνο μέχρι τη πληροφορία όπως θέλουμε. Σας ευχαριστούμε. Έχουμε δει και χειρότερα. Μάρκο Βάλλη. Ευχαριστώ πολύ και ευχαριστώ και τον Φίλιπ για τις στιγμές αναψυχής που μας προσέφερε. Ελπίζω αυτή η θερμή σχέση με τον Κούνορ να συνεχιστεί. Και πέραν αυτών των ευθύμων, ήθελα να πω ότι εμείς δεν έχουμε ιδιαίτερε ανησυχίες σε σχέση με αυτό το fast tracking, κυρίως ε, ή μόνο όσον αφορά αυτή την επισήμανση. η οποία θα μπορούσε να, να σημάνει κινδύνους ε, για σημαντικούς επενδυτές, αυτούς που έχουν ειδικό βάρος μεγάλο, που μπορούν να αποφασίζουν για ακόμη και ρηψοκίνδυνες επενδύσεις και μας απασχολούν ιδιαίτερα και τα υψηλά ποσοστά είτε που αφορούν ενδεχομένως ε, ε, στεξιδοτικά ταμεία, επενδυτικά ταμεία κτλ. Σε αυτό θέλουμε να δώσουμε ιδιαίτερη προσοχή μέσω των επενδύσεων μας. Κατά τα άλλα, όλη η πρόταση BRRD που βεβαίω θα μας υποχρεώσει σε μια ευρύτερη συζήτηση επόμενα, στους επόμενους μήνες, για μας σημαίνει αρκετές ακόμη επιφυλάξεις για λόγους πολιτικούς, διότι πιστεύουμε ότι ένα σύστημα εξυγίανσης σε σχέση με τα όσα έχουμε κάνει ε, από την προηγούμενη ήδη βουλευτική περίοδο για την προστασία των ε, μικροκαταθετών δεν ε, επαρκεί και γι' αυτό θα συνεχίσουμε να παρακολουθούμε τη συζήτηση και αυτές είναι οι παρατηρήσεις που μας ενδιαφέρουν. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ και πολύ σύντομα για να δώσω κάποια ναύσματα σε μια εις βάθος συζήτηση που πιστεύω θα προχωρήσει με τις συμβαστικές τροπολογίες του εισηγητή. Συνοψίζοντας και τις προτάσεις μας μέσα από τις τροπολογίες για την έκθεση αυτή, γιατί πρέπει να έχουμε σαφήσει τους εξής τρεις στόχους. Πρώτον, ότι θα πρέπει να δώσουμε σάρκα και οστά στην ε, BRRD, όσο και αν δεν συμμεριζόμαστε τις δομές, θα ήταν καλό να εξασφαλίσουμε κάποιες δυνατότητες προστασίας για τους θεσμικούς επενδυτές, μεγαλύτερη προστασία για τις ε, μη εξασφαλισμένες ε, ομολογίες, unsecured bonds και άλλες μορφές αποταμίεσης έτσι ώστε να προστατεύσουμε την αποτομίευση του Ευρωπαίου πολίτη. Δεύτερο θεμελιώδη ζήτημα, η διαφάνεια. Θέλουμε δηλαδή να έχουμε εργαλεία τα οποία, τα δευτερεύοντα εργαλεία, θα μπορεί να είναι ρηψοκίνδυνα, υψηλού κινδύνου για έναν ε, επενδυτή μικρού μεγέθους retail, αν και θα ήταν βέβαια ανόητο να πολλούνται τέτοια εργαλεία υψηλής διακινδυνεύσης ε, όπως οι μετοχές. Πώς όμως αυτό μπορούμε να κάνουμε προς το παρόν. Και έτσι θέλουμε στη MIFID 2 να προσαρτηθεί αυτό το νέο εργαλείο έστω και αν δεν ακολουθούμε την έννοια της ε, σκοπιμότητας που θα κάνει το καταλληλότερο αλλά το κριτήριο της καταλληλότητας δηλαδή ο κίνδυνος για τον μικρό αυτό επενδυτή θα είναι σχετικά υψηλός αλλά πάλι θα υπάρχει ένα ε, όριο καταλληλότητας σε σχέση με τον μεσολαβητή για τα όσα λένε οι σοσιαλιστές είναι σημαντικό η αρχική διάρκεια, η maturity δηλαδή των ομολόγων, να είναι τουλάχιστον ενός έτους. Για να διατηρηθεί η αναλογία και η συμμόρφωση με τις διατάξεις εκείνες οι οποίες εξασφαλίσουν περισσότερη δυνατότητα ε, ελέγχου παρακολούθηση από τους οργανισμούς. Περιμένουμε βεβαίως συγκεκριμένες προτάσεις πάνω στις οποίες θα μπορέσουμε να ε, εργαστούμε και να συνεργαστούμε με τον εισηγητή. Ευχαριστώ. Έχουμε εκπρόσωπο της Επιτροπής, ο κύριος Κούριν. Πολύ σύντομα παρακαλώ. Αλλά πιστεύω θα είναι χρήσιμο να σας ακούσουμε. Παρακαλώ. και εμείς αντιμετωπίζουμε πολύ θετικά τη δουλειά του Συμβουλίου και εδώ και αναμένουμε τον τριμερή διάλογο με ανυπομονησία. Θέλετε να τοποθετηθώ σε μερικές από τις προτινόμενες τροπολογίες και να σας πω την άποψη της Κομισιόν. Πρόεδρε. Να διευκρινίσω μερικά πράγματα για την πρότασή μας σε σχέση με τις τροπολογίες που έχουν ζητηθεί σε ό,τι αφορά την, αρχία, την αρχή της προτίμησης ε, των καταθετών. Η πρόταση που έχουμε υποβάλει έχει σχέση με μια πολύ συγκεκριμένη ταξινόμηση εφερεγγιότητας ε, που θέλουμε να εισάγουμε ε, για να γίνει πιο εύκολη η διάσωση με ιδίους πόρους με διαμέσα. Αυτό είναι απολύτως απαραίτητο προκειμένου να τηρούμε τα, τις προδιαγραφές TLAC ε, και να καταστεί πιο εύκολη η διάσωση. Δεν έχουμε μιλήσει για την προτίμηση των καταθετών, γιατί το ζήτημα αυτό είναι πολύ πιο περίπλοκο. Απαιτεί η εκτίμηση του δικτύπου, ε, στάθμιση των υπέρ και των κατά, γιατί όπως γνωρίζετε μερικά, μερικές τράπεζες και μερικά επιχειρηματικά μοντέλα βασίζονται σε καταθέσεις, σε εταιρικέ καταθέσεις για να πληρούν τις απαιτήσει ε, ε, ε TLAC. Τότε που υποβάλαμε την ε, πρόταση θέλαμε να προχωρήσουμε στην ε, ταξινόμηση και να υποβάλουμε μια άλλη πρόταση για το θέμα των ε, προτίμησης των καταθετών με άλλη σε κατοπινό χρόνο μεταγενέστερο στο χρονικό διάστημα. Τώρα, ε, η πρότασή μας αφορά την ταξινόμηση ε, της αφαιρεγγιότητας των τραπεζών. αυτό είναι το βασικό μας αντικείμενο. Τώρα, η προστασία των επενδύσεων είναι σε ένας παράγοντας. Υπάρχουν κανόνες στην οδηγία MIFID, και στόχος θα πρέπει να είναι αυτοί οι κανόνες να εφαρμόζονται, ε, να εφαρμοστούν αποτελεσματικά και όχι να τρομοποιηθούν. Νομίζω ότι οι κανόνες αυτοί είναι αρκετοί. Το πρόβλημα ενδεχομένως βρίσκεται στην εφαρμογή τους. Οπότε δεν βλέπουμε ισχυρά επιχειρήματα για να εντάξουμε τέτοιου διατάξεις. Εκτός από μία που είναι η αποκάλυψη των κινδύνων. Υπάρχει ήδη. Θα πρέπει οι κίνδυνοι, να είναι, οι κίνδυνοι που, που συνεπάγεται το μέσο που πληρεί τις από τις MREL και το πρότυπο TLAC, η κίνδυνη αυτοί θα πρέπει να είναι δεδομένη και γνωστή. Επίσης θέλουμε να συζητήσουμε το θέμα της ε, πατρόνικης ε, ε, χρειάζεται μια συνέχεια. Χρειάζεται μια συνέχεια. θέλουμε ε, να επιβαρηθούν οι τράπεζες που αυτή τη στιγμή πληρούν τις ελάχιστες απαιτήσεις MRL. Νομίζω ότι μπορούμε να το συζητήσουμε και να βρούμε μια λύση. Αυτά από πλευρά της Κομισιόν. Αν έχετε κάποιες πιο συγκεκριμένες ερωτήσεις, πολύ ευχαριστώ να απαντήσω. Thank you. Ευχαριστούμε. Τελικά σχόλια από τον ε, εισηγητή. Ευχαριστώ. Πολύ σύντομα. Πρώτον, στον ε, φίλο μου τον Φιλίπ, φίλος από τα παλιά. Δυστυχώς φαίνεται ότι οι σχέσεις μας έχουν αλλάξει. Έχει δίκιο όμως ότι στην πραγματικότητα εδώ ακολουθούμε το σκεπτικό της BRRD και το κάνουμε αυτό προκειμένου να συμπληρώσουμε την ε, ιεραρχία που προβλέπεται σε εκείνη την οδηγία. Δεύτερον, υπάρχει ε, συναντήληψη εδώ στην Επιτροπή ότι πρέπει να ε, ε αντιμετωπίσουμε το ζήτημα της, ε, της πατρογονικής ρήτρας. Ε, και εδώ πρέπει να ευθυγραμμιστούμε όσο το δυνατόν περισσότερο με το Συμβούλιο. Δεν υπάρχει κανένας λόγος ε, να, να βρίσκουμε διάφορες, τεχνικές μεθόδους ως αυτοσκοπό δηλαδή. Όσον αφορά αυτήν την νέα κατηγορία αφαιρεγγιότητας, αν κάποιο χρέος δεν έχει συγκεκριμένο ελάχιστη, ε, ε, συγκεκριμένη ελάχιστη διάρκεια, Προφανώ δεν πληρεί τα κριτήρια TILAC. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί στην περίπτωση ενός Μπέιλιν. Και αυτό αφορά και η πρόταση της Κομισιόν για αυτή την απέτηση ενός έτους. Προφανώς, αν δεν, αν δεν υπάρχει αυτό το κριτήριο, προφανώ δεν εκπληρώνονται τα κριτήρια TILAC. Παρ' όλα αυτά, αυτό δεν σημαίνει ότι δεν είναι κάτι, αυτό το χρέο δηλαδή, ε, που θα μπορούσε να χρησιμοποιηθεί στη διαδικασία ε, διάσωση με ίδια μέσα. Αυτά και σα ευχαριστώ για όλα τα σχόλια και προβλέπω στις από εδώ και πέρα συζητήσει αυτό το θέμα. Ε, ευχαριστώ. Θα προγραμματίσουμε να γίνει ψηφοφορία το συντομότερο δυνατό, λέει ο Πρόεδρος. Μια γενική δέσμευση να γίνει εντός του Οκτωβρίου, προκειμένου να ξεκινήσει το τότε δυνατό η, ο τριμμένος διάλογος, με την επιφύλαξη βεβαίως όλων των δικαιωμάτων των ε, μελών των, ε, του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου ε, και χωρίς να θέλουμε να προκαταλάβουμε τη στάση, προκαταλάβουμε τη στάση κανενός. Λοιπόν, και με αυτά μπορούμε να περάσουμε στις ψηφοφορίες. Πρώτον, θα ήθελα να κάνουμε μια δοκιμή. Ψηφίστε παρακαλώ ηλεκτρονικά για να δούμε αν λειτουργεί το σύστημα κανονικά. Uh, so, Ωραία, πέρας λοιπόν. Και ψηφίζουμε τη δική μου έκθεση, σχέδιο έκθεσης. Προσαρμογή διάφορων νομικών πράξεων οι οποίε προβλέπουν τη χρήση κανονιστική διαδικασία με έλεγχο στα άρθρα 290-291 της Συνθήκης για τη λειτουργία της Ευρωπαϊκής Ένωσης. Όπως ξέρετε, υιοθετήσαμε μια συγκεκριμένη διαδικασία. Πρόσθετες τροπολογίες δεν έχουμε λάβει. Ψερέφει όμως, πρέπει όμως να ψηφιστούν αυτές οι προτάσεις του εισηγητού. Τις έχουμε ομαδοποιήσει. Και έτσι ψηφίζουμε την ομάδα Α, υπέρ κατά, αποχές εγκρίνεται. Β υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Σ γάμα υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Δ δ, υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. Ή ε υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. F σιγματάφ υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. G ζ υπέρ κατά αποχές ε, εγκρίνεται H, ήτα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. I, θήτα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. J, ιότα υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. K, κάπα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. L, λάμδα, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. M, μη, υπέρ, κατά, αποχές, εγκρίνεται. Και τώρα, πρόταση της Επιτροπής όπως τροποποιήθηκε, ονομαστικά παρακαλώ, άρχεται η ψηφοφορία. Δεν Πέρας. 46 υπέρ. Μία ψήφος κατά, δύο αποχές. Σας ευχαριστώ. Και βεβαίως αναμένω ότι και στο μέλλον κάθε μου τροπολογία με τον ίδιο ενθουσιασμό και αμέριστη υποστήριξη θα εγκρίνεται τις τροπολογίες μου. Κύριος Λάμπερτς, θέλω πρέπει να διακόψω κύριε Πρόεδρε την ψηφοφορία και λυπούμε, αλλά μήπως θα μπορούσαμε να κάνουμε ομαδοποίηση των ομάδων για την επόμενη φορά. Να το σκεφτούμε λέει ο Πρόεδρος. Μια και αναφέρονταν σε διαφορετικά νομοθετήματα, θεωρήσαμε ότι ήταν σκοπιμότερο να τις ομαδοποιήσουμε κατά τον τρόπο που είδατε. Να λέτε και ευχαριστώ όμως που δεν σας βάλαμε να ψηφίσετε μία-μία τις τροπολογίες. Εντάξει, για την επόμενη φορά θα το λάβουμε υπόψη. Να κάνουμε ομάδες ομάδων. Ευχαριστώ και τώρα πάμε στο σχέδιο γνώμοδότησης της Μαρίζα Ματίας για την καταπολέμηση των ανισοτήτων ως μοχλό για την τόνωση της, δημοκρα... της θέσεων εργασίας και της ανάπτυξης υπέρ κατά αποχές. Εγκρίνεται. 42 υπέρ, κατά αποχές. Απερίφθη 45 υπέρ, κατά αποχές. Απερίφθη 46 υπέρ, κατά αποχές. Απερίφθη 47 υπέρ, κατά αποχές. Επαληθεύουμε. 47 άρχεται η ψηφοφορία. Πέρασε. Απερίφθη. 48 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Συμβαστική 4 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 55 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Συμβαστική 5 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 57 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. Συμβαστική 6 υπέρ. Κατά. Απόχες εγκρίνεται. 64 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 65 έχει αποσυρθεί. Συμβαστική 7 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 8 υπέρ συμβαστική κατά αποχές εγκρίνεται. Συμβαστική υπέρ 1 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται. 11 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 12 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 13 υπέρ κατά Επαλθεύω. άρχεται η ψηφοφορία πέρας απερίφθη 14 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 15 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 16 υπέρ κατά αποχές απερίφθη 17 υπέρ κατά αποχές απερίφθη συμβαστική 2 υπέρ κατά αποχές εγκρίνεται 24 υπέρ 24 υπέρ. Κατά. Αποχές απερίφθη. 27 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 28 υπέρ. Κατά. Αποχές εγκρίνεται. 29 υπέρ. Κατά. Απερίφθη νομίζω, αλλά σε παληθεύσουμε. Πέρας. Με όλα τα καλά σου λόγια σε καταψήφισε. 30 υπέρ κατά αποχές απερίφθη. 31 υπέρ κατά αποχές. 31. Επαληθεύουμε. Vote is Πέρας. Απεριφθεί. Το κείμενο αποστροποποιήθηκε ονομαστική ψηφοφορία παρακαλώ. Πέρας. 39 υπέρ, 9 κατά, μία αποχή. Συγχαρητήρια στον συγκεκριμένο. Και πέρα στη συνεδριάσεως προσεχή συνεδρίαση 9 Οκτωβρίου, 3 το απόγευμα, 10 Οκτωβρίου, πρωί και απόγευμα. Σας ευχαριστώ.